Äh, θα ήθελα να σας χαιρετήσω εγκαρδιότατα στη συνεδρίαση και να σας ανακοινώσω τις αλλαγές για την ημερησία διάταξη. Δυστυχώς ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρο δεν έχουν φτάσει ο χρόνο. αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω τη συνεδρίασή μας. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω τις αλλαγές που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Η πρώτη αλλαγή αφορά το σημείο 12 την νομοδότηση Beauty Coffer που θα το εξετάσουμε σαν 3α. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Μετά το σημείο 5, γνωμοδότηση Langen. Τη συζήτηση επί των τροπολογιών, η οποία θα γίνει σαν 3β. Η Επίτροπος Νέλη Κρούς θα έρθει κάπως αργότερα δηλαδή στις 4 το απόγευμα. Και θα έχουμε εξετάσει και τα σημεία 6 και 5. Για το σημείο 6 έχω να σας πω ότι η έκθεση Σόζα Βάγνερ, όπου θέλουμε να συζητήσουμε τι τροπολογίες, θα είναι το τελευταίο σημείο που θα εξετάσουμε την 21η Μαΐου. Μετά από στο σημείο 13. Έκθεση Τεγκράστα Καβάλιο είναι μια ανταλλαγή απόψεων που θα εξεταστεί σαν 11α μετά τις ψηφοφορίες αύριο. Η συνεδρίαση των συντονιστών δεν θα λάβει χώρα σήμερα, αλλά την τρίτη το πρωί, αύριο δηλαδή, μετά την ψηφοφορία και, τις και την συζήτηση εκθέσης Καρβάλιο, δηλαδή γύρω πολύ στις 11 και τέταρτο. Σημείο 14. Ο πρόεδρος Μπούσεκ θα σχολιάσει και την ε, επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να τη θεωρήσουμε εγκεκριμένη και να περάσουμε στο σημείο 3. Ε, Που είναι η έγκριση των πρακτικών Ε, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά, θα ήθελα να πράσουμε στο σημείο 4. Ist, die, uh, die, der Bericht... Στην ε, εξέταση της έκθεσης Beauty Cover Θα ήθελα να μας κάνει μια εισαγωγή εκείνος Beauty Cover αμέσως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης είναι σημαντικό για την εσωτερική αγορά και για οικονομικούς, ε, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Σε όλους αυτούς τους τομείς με προσφέρει πλεονεκτήματα η Ευρώπη. μπορεί να τηρήσει τη θέση της σαν μια περιοχή με μεγάλη εμπειρία τεχνολογική μόνο εάν εμείς ξέρουμε πώς θα ενδυναμώσουμε τους στόχους της πολιτικής μας. Και από την άλλη μεριά, η ευρωπαϊκή στόχοι τυποποίησης θα πρέπει βέβαια να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα και να αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις όπως είναι η ασφάλεια του εφοδότης με ενέργεια, οι κλιματολογικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Για να εκφράσουμε όλα αυτά στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής τυποποίησης θα πρέπει να έχουμε μια λύση που λαμβάνει υπόψη ευρύ φάσμα συμφερόντων και η τυποποίηση να μπορεί να καθοριστεί μέσα στα πλαίσια μιας διαφανούς διαδικασίας. Αυτά εισαγωγικά, ορισμένες πολύ γενικές παρατηρήσεις. Βασιζόμενος πάνω στις γενικές αυτές παρατηρήσεις, θα ήθελα να προτείνω για την γνωμοδότηση για την έκθεση που θα κάνει η Επιτροπή ΙΜΚΟ Ορισμένα θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να προτείνω τα σημεία ε, της ΠΟΕ, διαφάνειας, ανοιχτοσύνης, ε, ε, αποτελεσματικότητας και συνέπειας να συμπεριληφθούν στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τυποποίηση. Aus meiner Sicht äh, sehr wichtig, dass... Äh, Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι θα ήταν σωστό διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν κοινοφελή συμφέροντα να εμπλακούν πολύ περισσότερο στη διαδικασία καθορισμού της τυποποίησης αυτής. Παραδείγματο κάνει η NORMAPME, ε, η οργάνωση τυποποίησης των ΜΜΕ, η ΕΚΟΣ που εκπροσωπεί περιβαλλοντολογικά πρότυπα ή και άλλες οργανώσεις οι οποίες είτε από σκοπιάς καταναλωτών είτε από σκοπιά συνδικάτων και ασφάλειας ε, στον τόπο εργασίας εκπροσωπούν αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε. Θα ήταν καλό νομίζω η και αλλες οργανωσεις οι οποιες ειτε απο σκοπιας καταναλωτων ειτε απο σκοπια συνδικατων και ασφάλεια στον τοπο εργασιας εκπροσωπουν αυτο που θελουμε να διαθέσει πόρους ούτως ώστε οι ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης να υποστηριχτούν κατά την προσπάθειά τους καθορισμού προτύπων όπως αυτά που θέλει να έχει η Κομισιόν. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε ένα τμήμα των πόρων να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα για την υποστήριξη αυτών των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών στην διαδικασία τυποποίησης. Αυτά βέβαια μόνο εφόσον συγκεκριμένα πρότυπα εντάσσονται στις αρμοδιότητες αυτών των οργανώσεων. Πέραν αυτού, θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε την σημασία μας στη διαδικασία αντιποποίησης εφόσον ε, σε επίσημες αποφάσεις για τα λεγόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα να υπάρχει μία φωνή που να ακούγεται. Χωρίς αυτό να πλήξει τις σχέσεις ε, πλειοψηφίας, γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχει μια στάθμιση των ψήφων ε, στη διαδικασία αυτή η Γαλλία έχει παραδείγματο χάνει 10 ψήφου κλπ. Αλλά θα μπορούσαμε 5-10 ψήφου στη διαδικασία να τις δώσουμε στις οργανώσεις αυτές που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του πολίτη. Και έτσι θα μπορούσαμε να λάβουν υπόψη μας τα συμφέροντα διαφορών ενδιαφερομένων. Τέλος, θα πρέπει τα πρότυπα αυτά να είναι προσιτά Τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκά σε διάφορε από τι διαδικασίε που συζητάμε. Το κόστο επίση είναι αρκετά υψηλό, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ε, διεθνείς οργανώσεις τυποποίησης θα πρέπει να προσφέρουν ιδίως στις ΜΜΕ σειρά προτύπων και τα πρότυπα αυτά πρέπει επίσης να απλουστεύονται εφόσον μειωθεί η αναφορά που γίνεται σε άλλα ε, πρότυπα και σε άλλους τύπους. Αυτό θα διευκολύσει νομίζω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση τους αυτών των προτύπων τυποποίησης. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει καλός συντονισμός των δικών μας προτύπων τύπων με την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να αναπτυχθούν δραστηριότητες για να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και ακόμα και στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου να τονίσουμε το θέμα αυτό των προτύπων. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θα πρέπει να εξτάσουμε το θέμα του διεθνούς συντονισμού σε περίπτωση τυποποίησης. Δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό γιατί ανταγωνισμός προτύπων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη δεσμολογικά εμπόδια και ιδίως όσον αφορά τις σύγχρονες καινούριε τεχνολογίες θα μπορούσε έτσι να πανεμποδιστεί η εξέλιξη των αγορών. Και γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε ούτως ώστε το γλυγορότερο δυνατόν να οδηγηθούμε σε μια επιτάχυνση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τον Διατλαντικό διάλογο και το έργο του Διατλαντικού Συμβουλίου Οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποιος ε, Ευχαριστώ κύριε Βητυχόφερ. πώς θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας του. Αυτό το θέμα των πρωτοτυπών είναι ουσιαστικότατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία αρχή τυποποίησης και όποιος θέλει να προστατεύσει τους ε, καταναλωτές Βλέπετε ότι με τον τρόπο αυτό επιτυχάνεται μεγάλη επιτυχία και μπορέσαμε πολλά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα να περάσουν σαν διεθνή πρότυπα. Έχω παραδείγμα χάρη το τον κανονισμό REACH στην χημική βιομηχανία που πολλοί μας ακολούθησαν σε αυτό. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν. Αλλά όσον αφορά τα πρότυπα τεχνικά και οικονομικά για τα οποία είχαμε επιτυχία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα πρότυπα που δεν σχετίζονται άμεσα με την χώρα. Αναφερθήκατε στα περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Η προστασία της ζωής μας, ε, του πλαισίου ζωής όσον αφορά τις περιβαλλοντικές Τα Θα με υγειονομικά πρότυπα να έχουμε κοινωνικά, πολιτιστικά. Όσον αφορά αυτά τα πρότυπα που εξέρχονται της αγοράς, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα επιβάλλουμε. Θα ήθελα εδώ να σας ε, υποδείξω την αποτυχία, τέλο κατά το ίμιση αποτυχία της διάσκεψης κορυφής της Κοπενχάγης, όπου οι οργανισμοί που θέλαν να ορίσουν τα πρότυπα αυτά δεν κατάφεραν να παίξουν το ρόλο του καλού παραδείγματος και να παρασύρουν το υπόλοιπο του κόσμου μαζί τους. Απέτυχαν λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε τα πρότυπα αυτά. το 4x20, ορισμένοι λένε 4x30. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εάν εμείς επιβάλλουμε αυτά τα περιβαλλοντικά πρότυπα και έτσι πλήττουμε σκληρά τις δικές του βιομηχανίες σε σχέση με άλλες χώρες, ε, αναδυόμενες αλλά και τη ΣΥΠΑ και άλλες, που δεν εφαρμόζουν παρόμοια πρότυπα. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Ορισμένοι, όπως η γαλλική κυβέρνηση, αλλά και τα κύρια κόμματα της αριστεράς στη Γαλλία, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φόρος του άνθρακα στα σύνορα για να επαναφερθεί έτσι η ισότητα στον ανταγωνισμό και γενικά ρωτάω τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε όταν υπάρχει σύγκρουση των προτύπων μεταξύ των ε, οικονομικών προτύπων και των προτύπων εκτός αγοράς για να βρεθεί μία λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μόνο εθελοντική, παραδειγματική στάση, όπως είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή καταγράφει τα όρια. Γιατί δεν μας ακολουθούν για πολλά θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια χωρίς να κάνουμε τίποτα, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια μάχη προτύπων σε διεθνώς επίπεδο. Και γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε, να διευκρινίσουμε ε, τι πρέπει να γίνει και να μας πει ο εισηγητής ποια είναι η άποψή του από αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα θέματα που θίξατε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά για μας γιατί η τυποποίηση θα παίζει και στο μέλλον μια, ένα σημαντικό ρόλο. Ο Επίτροπος Φερχόγγεν είχε πει ότι θα πρέπει να έχουμε λιγότερη τεχνική νομοθεσία και η τυποποίηση να αναθεθεί στα αρμόδια βήματα και να υπάρχουν εκεί νέοι τομείς αρμοδιότητας. Πάλι λοιπόν πρόκειται εδώ για την βασική αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνησης πού θέλουμε αμοιβαία αναγνώριση και πού θέλουμε εναρμόνιση. Αυτά τα δύο επίπεδα θα πρέπει να τα εξετάσουμε εις βάθος, γιατί και στα 27 κράτη-μέλη έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε την τυποποίηση και μάλλον θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αναγνώριση. αναγνώρισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε παρόμοια επίπεδα, η τυποποίηση είναι πραγματικά, η εναρμόνιση συγγνώμη είναι πραγματικά μια πρόκληση. Και στην οικονομία έχουμε τα διεθνή πρότυπα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα πρέπει να φροντίσουμε στην εσωτερική μας αγορά ποια είναι τα πρότυπα που χρειαζόμαστε, πόσα τυποποίηση χρειαζόμαστε και το θέμα που έδειξε ο κύριος Βιτικόφερ του κόστους και της χρηματοδότησης του συστήματος παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο. Δεν βλέπω κανένας άλλος να θέλει το λόγο, οπότε θα ήθελα ίσως η Κομισιόν να τοποθετηθεί. Ο κύριος Ντύρσε είναι εδώ παρόν και αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Βέβαια τώρα που να τρέψαμε την Ευρωπαϊκή, την ημερησία διάταξη είναι λογικό ότι δεν είναι παρόν. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε Η προσεχή συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότηση είναι 23 Ιουνίου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 24 ε, Ιουνίου, 5 το απόγευμα. Η συζήτηση των τροπολογιών αυτών και η ψηφοφορία θα γίνει 13 Ιουλίου και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ η ψηφοφορία προβλέπεται για 2 Σεπτεμβρίου 2010 και γι' αυτό η, ομολ... η Ολομέλεια θα το εξετάσει είτε στη δεύτερη σύνοδο του Σεπτεμβρίου είτε στην πρώτη του Οκτωβρίου. Εάν συμφωνείτε όλοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μπιουτικόφερ για να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και τον κύριο Βέμπερ για τα σχόλια που εκφράσατε και τις ε, σκέψη σα, Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Επανέρχομαι σε δύο-τρία ε, σχόλια που έγιναν. Δεν είμαι βέβαιος εάν η διεύρυνση του θέματος, όπως προτείνει ο κ. Βέμπερ, μπορεί να ενταχθεί, να υπαχθεί σε τούτη εδώ την προσπάθεια. Εκτιμώ την σημασία των προτύπων. Ίσως βέβαια να μην κατανόησα καλά τι είπε ο κύριος Βέμπερ, τουλάχιστον πάντως αυτό άκουσα. Δεν θεωρώ πάντως την σημασία των προτύπων σαν κάτι το οποίο είναι μια επιβάρυνση ή μια δυσχέρεια για τη βιομηχανία. Εγώ βρίσκω ότι είναι μάλλον ευκαιρία για την βιομηχανία και ανεξάρτητα τώρα από την ευρύτερη συζήτηση του λεγόμενου carbon leakage οι έρευνες που γίνονται πρόσφατα και που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι τόσο δύσκολο όσο το έχουν εμφανίσει ορισμένες πλευρές. Εάν πάντως δεν περιοριστούμε μοναχά στην ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά για παράδειγμα λάβουμε και υποσημείωση τον φιλόδοξο τρόπο με τον οποίο ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες προωθούν τεχνολογικές καινοτομίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, τότε νομίζω ότι οφείλουμε να αποτιμήσουμε πραγματικό φόρο τιμής ή στις προσπάθειες των χωρών αυτών που δεν περιμένουν να τρέχουν από πίσω μας αλλά προχωρούν και δείχνουν τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν είμαστε πλέον σε κατάσταση όπου μπορούμε να σκεφτούμε αν θέλουμε να είμαστε πρότυπο για άλλους. Οι Κινέζοι, για παράδειγμα, δεν περιμένουν πλέον από την Ευρώπη να παίξει ρόλο πρότυπου. Αντίθετα προσπαθούν να μας ξεπεράσουν ε, στην έρευνα και χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Έτσι λοιπόν ε, θα θεωρούσα ότι από άποψη βιομηχανικής πολιτικής είναι επικίνδυνο να διαδίδεται η άποψη ότι ίσως πρέπει να κάνουμε την χάρη στην βιομηχανία, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εισαγωγή κοινών προτύπων, να βαδίσουμε πολύ προσεκτικά. Αντίθετα, νομίζω με την ανάπτυξη κοινών προτύπων πρέπει να συμβάλλουμε ώστε ο, ο, ρυθμός, η επιτάχυνση των, ε, της χρήσης των τεχνολογιών αυτών να είναι μεγαλύτερος. Ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Ακολουθεί το θέμα των επιδόσεων από την άποψη των εκπομπών καυσαερίων των ελαφρών φορτηγών οχημάτων. Ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην φάση συζητήσεως των τροπολογιών, εκ των οποίων υπάρχουν συνολικά 219, οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε 18 επιμέρους παραγράφους. Η πρώτη τροπολογία αναφέρεται στην νομική βάση. Αν δηλαδή πρέπει να πάρουμε ως επιπρόσθετη νομική βάση και την ε, και το άθρο της ενιαίας αγοράς. Υπάρχει όμως ήδη γνωμοδότηση σχετικά με τα επιπαιδευτικά αυτοκίνητα που λέει πως όχι. Δεύτερο μεγάλο σύνολο θεμάτων είναι των βραχυπρόθεσμων τιμών στόχων και σε ό,τι αφορά το ύψος αλλά και σε ό,τι αφορά την διάρκεια. Σε ό,τι αφορά το ύψος υπάρχουν προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 175. Έχουν γίνει και προτάσεις χαμηλότερες από την κυρία Χαρμς, την κυρία Χολ, Βάγνερ, Τόμψον και ορισμένους άλλους, 165 και 160 δηλαδή, εγώ προτείνω πάντως, έχοντας γνώση της πραγματικότητας, να ε, παραμείνουμε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τα 175 γραμμάρια. Η δεύτερη τιμή είναι η μακροπρόθεσμη. σε σχέση δηλαδή με την θέση σε ισχύ αλλά και τη μακροπρόθεσμη τιμή. Ο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 135 γραμμάρια με αυξήσεις στα 160, ελαφρές αυξήσεις στα 150, μειώσεις στα 125, 130, 145, με τροποποίηση και του αριθμού ετών 135 στο 2025 αντί για το 2020 και σταδιακά. Εγώ είπα ότι θα αποσύρω την πρόταση αυτή και θα προτείνω μια συμβαστική τροπολογία η οποία θα βρίσκεται στη μέση περίπου, στα 150 δηλαδή γραμμάρια και ταυτίζεται με αυτήν που έχει περιγράψει στην εκθεσή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος. 150. Αυτός ο στόχος είναι αρκετά φιλόδοξος και απαιτεί αρκετές προσπάθειες από τη βιομηχανία και τα θέματα που τίθεται φαίνονται να είναι ε, τα ερωτήματα που τίθεται να είναι σκόπιμα. Τώρα, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Εδώ υπάρχουν δύο τροπολογίε που αναφέρονται στα οχήματα κατηγορία μη 2 και νη 2, για να περιληφθούν δηλαδή και αυτά. Η ε, Κομισιόν αναφέρεται μονάχα στα νη 1 και εγώ θα ήθελα να περιστούμε στην πρόταση τη Κομισιόν. Υπάρχουν τώρα και συμπληρώσει των ορισμών το ίχνος άνθρακος ολόκληρου του χήματος κτλ. Όλα αυτά τα δέχομαι. Έκτο, το είναι το θέμα πότε θα αρχίσει. Phase in δηλαδή στα αγγλικά και εδώ τίθεται το ερώτημα πότε αρχίζει η ισχύς του κανονισμού αυτού. Εδώ έχουν γίνει προτάσεις για ε, σταδιακή εφαρμογή για το διοξείδιο του άνθρακος των φορτηγών οχημάτων, αλλά υπάρχουν και πιο λεπτομερείς που ε, προτείνουν σταδιακότερη εφαρμογή από την κυρία Τικάου δηλαδή, την κυρία Χάμς επίσης, η οποία δεν προβλέπει face-in και θέλει να εφαρμοστούν οι τιμές χωρίς face-in όπως είπα, η δική μου πρόταση είναι από το πλήθος αυτών των προτάσεων τροπολογιών να λάβουμε ως ημερομηνία αρχής να την αναβάλουμε αυτήν στην 1η Ιανουαρίου 2015. Και η σταδιακή προσαρμογή της ε, ε, Κομισιόν να συμπληρωθεί για τον πρώτο χρόνο με το 65% και από το 2016 να περιληφθούν τα πλήρη οχήματα, δηλαδή και με τις υπερκατασκευές. Μετά έχουμε, είναι περίπου τέλος πάντων η μέση οδός όλων των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Αν βέβαια όλοι επιμείνουν και καλά να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες τους, δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Επτά έχουμε το θέμα των super credits. Εδώ ζητείται από διαγραφή μέχρι ενίσχυση. Τα πάντα δηλαδή προτείνονται ως τροπολογίες. Και εδώ πάλι λαμβάνοντα υπόψη και του κανόνε του διοξιδίου του άνθρακο για τα φορτηγά οχήματα, θα προτείνω μια αλλαγή όπως αυτοί που προτείνουν Ρίμπικ, ε, Χατζημαρκάκης, Βάλιαν κλπ. Δηλαδή να μην ληφθούν ως αρχή τα 50 γραμμάρια, αλλά τα 50% της καθορισμένης ε, τιμής στόχου. Μου φαίνεται πιο σωστό αυτό, γιατί τα 50 γραμμάρια βέβαια δεν μπορεί να περάσει από τα φορτηγά στην κατηγορία των μικρότερων οχημάτων. Και μία πάλι εκεί σταδιακή προσαρμογή του υπολογισμού αυτών των ιδιαίτερα φιλικών στο περιβάλλον οχημάτων, 3,5 για το 2015 και μετά μέχρι 1,5 το 2018, δηλαδή κάπως πιο γενναιόδωρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε και τροπολογίες για το monitoring, monitoring συγγνώμη για την παρακολούθηση της εφαρμογής, που νομίζω ότι είναι περισσότερο ε, προσαρμογές των διατυπώσεων, των φαστικών διατυπώσεων. Τώρα, οι κυρώσεις, πρόστιμα κλπ. Εδώ προτείνω την ε, υπαριθμόν 4 συμβιβαστική, όλα λοιπόν θα αρχίσουν το 2015, αν αρχίσει από τότε να ισχύει ο κανονισμός, και το πιο σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 120 ευρώ εφόσον υπερβαίνεται η τιμή κατά 3 γραμμάρια, ανά τρία γραμμάρια δηλαδή υπέρβαση, όπως έχει γίνει και για τα φορτικά 2015-2019 και από το 2020 και μετά ακριβώς 95 ευρώ θέλουμε εμείς, δηλαδή λίγο λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πάλι ανταποκρίνεται, αν τα βλέπω σωστά, στις προτάσεις που κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και τώρα ερχόμαστε και στις προθεσμίες δημοσιεύσεων. Αναβολή κατά ένα έτος. Ε, Ρίμπικ Μαρινέσκου, Χατζημαρακάκης και Βαλιάρ. Συμφωνώ με αυτήν. Επίσης το θέμα των εξαιρέσεων. Αύξηση των τιμών ε, στόχων για μικρούς κατασκευαστές. 2020 προτείνει η Επιτροπή. Η τροπολογία της κυρίας Τικάου προτείνει 30.000, η δική μου πρόταση λέει 25.000 και νομίζω ότι θα τα βρούμε γιατί δεν είναι και ιδεολογικό το θέμα πώς θα διαμορφωθούν δηλαδή οι πλειοψηφίες. Τώρα, οι οικολογικές καινοτομίες. Εδώ ζητεί διαγραφή η κυρία Χάρμς. Χατζημαρκάκης, Βαλαιάν, Ρίβιχ, Μαρινέσκου, Τικάου. Θέλουν προσαρμογή στους κανονισμούς για τα φορτηγά αυτοκίνητα και η κυρία Τικάου προτείνει αύξηση από τα 7 στα 10 γραμμάρια. Εδώ είναι τεχνικό μάλλον το θέμα και σχετικά επίσης με το πώς όταν δηλαδή οι υπερκατασκευές αυτές δεν γίνονται μέσα στην ε, σύραγγα, ε, την αεροδυναμική σύραγγα, δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή εκεί, να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ρωστικότητα. Δεν μπορούν να σχεδιαστούν μέσα στην αεροδυναμική σύραγγα. Έρχεται τώρα το επόμενο κρίσιμο θέμα, οι ε, συσκευές περιορισμού της ταχύτητας. Εδώ υπάρχει πλήθος τροπολογιών. Από την αιτιολογική σκέψη 24 που ζητείται διαγραφή και συμπερίληψη νέας ε, αιτιολογικής σκέψης για την θετική ε, απόδοση των συσκευών περιορισμού της ταχύτητας Υπάρχουν και άλλε τροπολογίε οι οποίε υποστηρίζουν τη δική μου στάση και προέρχονται από διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Η κυρία Χάρμ, Βαν Μπρέμπτ και Κότεν θέλουν επέκταση του πεδίου εφαρμογή στην οδηγία 92-6 της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία σειρά από συναδέλφους κυρίως των Πρασίνων αλλά και κύριος Κότερ ζητούν νέο άρθρο 5α με διαφορετικά όρια. 120 χιλιόμετρα, κ. Σκότερ 110 και άλλοι, ε, ορισμένοι άλλοι βουλευτές, και Χάρμς και άλλοι 100, 100 χιλιόμετρα χιλιόμετρα. Που θα καθορίζουν, και άλλοι που θα λένε ότι θα καθορίζουν οι χώρες μέλη. Εκεί θα γίνει μαχητική ψηφοφορία. Την άποψή μου την έχω διατυπώσει στις τροπολογίες. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε υποχρεωτικό ούτε και σωστό. Γιατί το θέμα των ε, περιορισμών των ορίων ταχύτητος είναι θέμα των χωρών μελών. Έχουμε τώρα την αυτόνομη αύξηση μάζας. Πάλι εδώ υπάρχουν ορισμένε τροπολογίες Ρόμπι Χατζημαρκάκη Σαρτόρι, ε, Τικάου και ενδεχομένως αυτές να ψηφιστούν από πλειοψηφία. Εδώ η συμβιβαστική τροπολογία φέρει τον αριθμό 6. 6 λοιπόν. Που τάσεται υπέρ της διαγραφής. Τώρα, η συμπερίληψη της ε, κατηγορίας είναι δύο οχημάτων. Ε, Συμβαστική τροπολογία 5 που είναι άρθρο πολύ ευρύ αυτό με έναν αριθμό θεμάτων στη συμβαστική αυτή τροπολογία που πάλι στην ουσία προσανατολίζονται σε μια μέση οδό. Έχουμε και εναλλακτικές ε, τροπολογίες, έχουμε ε, εναλλακτικές μάλλον τιμές που προτείνει ο κ. Σοντή, έχουμε τα οχήματα με υπερκατασκευές διαφορετικών χρήσεων εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερη η μεθοδολογία. Όλες οι τροπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ο κ. Σωτής ζητεί διαγραφή. Οι άλλες τροπολογίες πάντως, όπως είπα, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2011 να προτείνει νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος. Και το τελευταίο είναι η διαβίβαση των δεδομένων. Αντί το 2011 προτείνεται εδώ το 2013. και την διαβίβαση των δεδομένων εκπομπών μαζί και με τις οικολογικές καινοτομίες. Δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται εκεί λοιπόν. Έχω λοιπόν προτείνει έξι συμβαστικές τροπολογίες που θα ήθελα, εάν δεν έχουν ήδη υποβληθεί, να υποβληθούν αμέσως μετά την συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την περαιτέρω εξέλιξη, έχει γίνει συζήτηση με τον κ. Κάλαχαν σχετικά με την οριοθέτηση του περιεχομένου. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα συζητήσουν ακόμα οι πρόεδροι των επιτροπών σχετικά με το ποιε είναι οι αποκλειστικέ αρμοδιότητε τη Επιτροπή Βιομηχανία. Έχουμε πάντω συμφωνήσει ότι ο καθένα θα κάνει την έκθεσή του πρώτα και μετά θα διαβουλευτούμε από κοινού για τα πράγματα που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα συζητήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πάντως, μέχρι τώρα υπάρχει σχετικά μεγάλη συμφωνία με τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχω προτείνει εγώ ίδιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βέρνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε από μία πρώτη ανάγνωση των τροπολογιών στην έκθεση του συναδέλφου Λάγγεν διαπιστώνουμε ότι υπέστησε περισσότερες υπάρχει ε, ένας κοινός παρονομαστής έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι στόχοι για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στα ελαφρά οχήματα. Εάν έχουμε μακροχρόνιους στόχους, ε, αυτοί οι στόχοι δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Και εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και πολλές φορές είπα για ποιο λόγο προβάλλω αυτές τις απαιτήσει λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα επαγγελματικά οχήματα αποτελούν μία αγορά που δεν είναι τόσο δυναμική σε σχέση με τα επιβατικά τα τελευταία δέκα χρόνια, πέρα από τον κύκλο παραγωγής που είναι μακρύτερος λαμβάνοντας υπόψη τα 35 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα που προτάθηκαν από την Επιτροπή, που σημαίνουν μεγάλες προσπάθειες από τον τομέα της βιομηχανίας, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στην βιομηχανία για να προσαρμοστεί γι' αυτό. Υπέβαλα μία τροπολογία όπου προτείνω να ε, προβάλλουμε μία παράταση από το 2020 στο 2025 για την ισχύ αυτών των τιμών. Επίσης, 160 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο θα ήταν ε, ένας εφικτός στόχος. Η Επιτροπή θα πρέπει μέχρι το 2011 να μας μιλήσει για τις διαδικασίες και για τον αριθμό των ε, οχημάτων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Βρισκόμαστε σε μια, σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης, κρίση στην απασχόληση, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ορίζουμε αυστηρά όρια. Έχω υποβάλει λοιπόν ορισμένες τροπολογίες γιατί θεωρώ ότι τα 135 γραμμάρια θα πρέπει να είναι 125. 125 γραμμάρια δηλαδή ανά χιλιόμετρο. Δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνολογία είναι έτοιμη να δεχτεί αυτές τις παραμέτρους. Πρόκειται για ένα επαχθές εγχείρημα το οποίο θα είχε επιπτώσει στην απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λάγκεν για την εργασία του επί του θέματος και για μια εκτενή ε, παρουσίαση της όλης ε, πρότασης. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα που δεν αναφέρθηκαν, αλλά επί των οποίων συμφωνούμε. Το ένα είναι το επιχείρημα της βιομηχανίας, ότι είναι ένας δυσλειτουργικός πλέον τομέας και αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν εφήγει αφορά τον υπολογισμό όπως ισχύει για τα super credits, αλλά μιλάμε για αρνητικά super credits, δηλαδή τα οχήματα που έχουν υψηλές εκπομπές, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε τα super credits και το αντεπιχείρημα είναι ότι αποτελεί δέλεαρ για τους κατασκευαστές έτσι ώστε να κατασκευάσουν οχήματα με υψηλέ εκπομπές. Επειδή ακριβώς παίρνουν super credits για τα οχήματα χαμηλών εκπομπών. Επειδή υπάρχει ένα χάσμα εδώ μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να προβάλλει καινοτομίε. Και αν δούμε τι συνέβη στα αυτοκίνητα, είδαμε ότι η βιομηχανία κινήθηκε πιο γρήγορα από ό,τι όριζε η νομοθεσία CARS και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και καθημερινά βλέπουμε ότι τα κοινά επιβατικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν μια κανονική τεχνολογία, την υπάρχουσα δηλαδή, έχουν ε, χαμηλότερες εκπομπές. Έχουμε, ας πούμε, ένα από τα τελευταία μοντέλα της Skoda. Νομίζω, λοιπόν, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καινοτομία, γιατί εκεί έγκυται το μέλλον για την απασχόληση. Είπα έχουν μείωση 5% στις εκπομπές. Άρα εμείς δεν θα θέλαμε να υπολοιπόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να μην αφήσουμε τη βιομηχανία να, να κινηθεί όπως κινείται τώρα. Υπάρχει το δέλεαρ να κινηθεί όπως κινείται μέχρι τώρα. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε με το τμήμα της βιομηχανίας που βρίσκεται πολύ πίσω, δηλαδή την καινοτομία. Επίσης, μπορούμε να μιλάμε για super credits για 50 γραμμάρια γιατί αυτά τα super credits για τα 50 γραμμάρια προωθούν τις νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα χαμηλών εκπομπών. Γι' αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε μία πρημοδότηση έτσι ώστε να έχουν κίνητρα. Ως προς τη νομική βάση, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, άρα η συνιστόσα του περιβάλλοντος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να δεχτούμε τους χαμηλότερους αριθμούς. Θα μιλήσω για αυτά τα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι οι εκπομπές είναι ο καθοριστικός παράγοντας και οι μικρές επιχειρήσεις μας ζητούν να έχουμε αυστηρούς στόχους επ' Και τα συνδικάτα, η συνομοσπονδία είναι απόλυτα σαφής. Θέλει χαμηλότερες εκπομπές και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μέσα σε αυτές τις τροπολογίες. Αυτό αφορά και τις κυρώσεις 120 γραμμάρια είναι ένα επίπεδο το οποίο δίνει κίνητρα στη βιομηχανία να κάνει κάτι διαφορετικό. Παρά να θεωρήσει ότι οχλείται κατά κάποιο τρόπο, αν συνεχίσει ως έχει. Τώρα, κατά πόσο θα είναι κάποιο καταποκοπή ποσό αυτό το πρόστιμο, αυτό μπορεί να συζητηθεί. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μακριά. Ο κύριος Λάγκεν ε, μίλησε για τροπολογίες συμβιβασμού. Δεν είδα το κείμενο. Ελπίζω να είναι διαθέσιμο, αλλά θα ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε με τους σκιώδεις και ίσως ο κύριος ε, Λάγκεν μπορεί να μας διευκολύνει ως προς αυτό. Έτσι ώστε φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο κύριος Ζαντό. Μετά την ε, παρέμβαση της κυρίας Χολ, συμφωνώ επί της ουσίας γιατί προβλέπεται μία συνεδρία μεταξύ εισηγητή και σκιωδών σε σχέση με τα ποσοστά. Πέρα από τα τεχνικά καθαρά θέματα, σήμερα αντιμετωπίζουμε μία συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση, όπως και στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας και δεν έχουμε παρά δύο επιλογές. Καταρχήν, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις όπως το ζητούν. Και μιλώ για τις περισσότερες, τις μεγαλύτερες. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο, να αποστασιοποιηθούμε κάπως, διότι Παραδείγματος χάρη στο Κογκρέσο της ΗΠΑ είχε ζητηθεί λιγότερος παρεμβατισμός από το κράτος, ιδιαίτερα για την General Motors και βλέπουμε σήμερα την κατάσταση. Η General Motors δεν έχει καμία κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο. Παρόλο που είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες, υπάρχει και μία άλλη επιλογή. Να θεωρήσουμε ότι με βάση τις δεσμεύσεις ως προς μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Νότιο Κορέα όταν αλλάξουν οι τιμές ενέργειας και όταν ανέβουν πάλι θα βρεθούμε με βιομηχανίες και καταναλωτές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Άρα ο ρόλος του Κοινοβουλίου και των πολιτικών είναι οι επιχειρήσεις να έχουν ένα πιο μακρόπνο και φιλόδοξο ορίζοντα. Και νομίζω ότι σήμερα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί μεταξύ των δύο. Δηλαδή, ή θα ακολουθήσουμε τις επιχειρήσεις, είτε θα επιβάλλουμε μία πιο φιλόδοξη ρύθμιση. Εδώ και δύο χρόνια είχαμε μία συζήτηση για τα επιβατικά και, είπαμε ότι, και είδαμε ότι αυτό που ήταν αδύνατον τότε για τη βιομηχανία δεν είναι τώρα. Κινείται πολύ πιο γρήγορα στα πλαίσια του εφικτού. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία για τα ελαφρά οχήματα να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Και θα πρέπει να μιλάμε για 160 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα για το 2014 και έναν πιο μακρόπνο στόχο για το 2020. Δηλαδή να προβάλλουμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες ε, οι οποίες σέβονται τις κλιματικές αλλαγές αλλά και τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που προελέχθησαν και γνωρίζω ότι ο συγητής αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε και τη γνωμοδότηση της Ένδυ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Χολ για αυτά που είπατε για την καινοτομία. Οι τροπολογίες μου είναι οι 80 και οι 85 σε σχέση με τα όρια ταχύτητας και διαξίδιο του άνθρακα, διότι συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν με την αύξηση του, των καυσίμων, του κόστου των καυσίμων. Όταν μιλώ με τους υπεύθυνους των ελαφρών φορτηγών, των φορτηγών, βλέπω ότι ασχολούνται ιδιαίτερα με την αύξηση των τιμών. Έγιναν συζητήσεις και πολλοί μου λένε ότι αν υπήρχε όριο ταχύτητας, τότε θα μειωνόταν το κόστος και θα είχα ένα ευεργέτημα. Άρα τα όρια ταχύτητας είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αλλά αν υπήρχε ταχυγράφος ή κάποια άλλη καινοτομία για την μείωση ε, κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, τότε θα μπορούσε να γίνει και αυτός ο υπολογισμός των εκπομπών. Και έτσι ο αγοραστής ενθαρρύνεται σε αυτή την περίπτωση. Τη στιγμή που υπάρχει ένας ε, ταχυγράφος ε, που δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά ο κατασκευαστής βλέπει ότι υπάρχει ευεργέτημα και γι' αυτό προβάλλει αυτές τις καινοτομίες. Ίσως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. κύριε Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή και τον ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι μας έδωσε μία συνολική εικόνα. Πρόκειται για ένα φάκελο ο οποίος είναι καθοριστικός για να αποφανθούμε και βεβαίως θα αποφανθεί και η ΕΜΒΗ. Θα ήθελα να υποβάλω ένα τεχνικό ερώτημα προς τον εισηγητή γιατί μιλάμε για συμβιβαστικές τροπολογίες. Θεωρώ ότι μιλάτε για αυτή την Επιτροπή αλλά δεν είχαμε την ε, ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με όλες τις πολιτικές ομάδες της ΕΜΒΗ. Με βάση τώρα αυτά που είπε η, κυρία Χάλ και ο κύριος Ζαντό, πολύ συχνά όταν μιλάμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη, μας λένε ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στις νέες τεχνολογίες, διότι θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε φιλόδοξους στόχους και συνειδητοποιώ ότι αρχίζουμε να φοβόμαστε όταν ε, θέλουμε να φανούμε φιλόδοξοι για να επιβάλλουμε ρυθμίσεις στη βιομηχανία. Εγώ έχω διατυπώσει φιλόδοξους στόχους, αλλά φοβάμαι τις συμβιβαστικές που θα αποδυναμώσουν την πρόταση της Επιτροπής. Ξέρω ότι είναι ρεαλιστική η Επιτροπή γενικά και οι προτάσεις της Επιτροπής ε, συχνά αποτελούν κάτι το ε, εφικτό για τη βιομηχανία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Από τη δική μου πλευρά πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε προτάσεις που αποδυναμώνουν το κείμενο της Επιτροπής. Υποστηρίζω τη θέση του εισηγητή για τον περιορισμό ταχύτητας και για το μηχάνημα αυτό που θα ανοιχνεύει την ταχύτητα. Εγώ έδωσα μεγάλη μάχη και γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια πολύ καλή πρόταση και σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες. Σύντομη γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Uh, thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν για αυτή την πολύ καλή σύνοψη της πληθώρας αυτής τροπολογιών που είναι αρκετά ε, περίπλοκες. Θα ήθελα να δω τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού, να δω, να δω πού έγκυται ο συμβιασμός μεταξύ όλων αυτών των αριθμητικών στοιχείων και ημερομηνιών. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε ως προς το συνολικό πακέτο. Δέχομαι αυτά που είπαν πολλοί ομιλητές, χρειαζόμαστε φιλόδοξες προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της βιομηχανίας. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις με τη, την ολοένα ε, και μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο όγκο ε, εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, γι' αυτό πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να έχουμε βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους. Και αυτά τα στοιχεία στην πρόταση της Κομισιόν βασίζονται σε μια μελέτη αντικτύπου μετά από διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και θεωρήσαμε ότι ήταν ε, ρεαλιστικά στοιχεία. Όπως ανέφεραν και άλλοι, και όπω αναφέρεται και στο έγγραφο τη Επιτροπής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, η καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Μόνο όταν έχουμε φιλόδοξου στόχου για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέσω νέων τεχνολογιών μπορούμε να έχουμε μια καινοτόμο τεχνολογία. Μόνο αν έχουμε ρύθμιση μπορούμε να καινοτομήσουμε. Αυτά είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας. Ένας ε, τομέα που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι η χρήση των super credits στην πρότασή μας θεωρήσαμε ότι τα super credits πρέπει να ισχύουν ε, αν υπήρχαν οχήματα που εκπέμπουν κάτω από 50 γραμμάρια στην αγορά. Γιατί αν θέλουμε να υπάρχουν ηλεκτρικά ελαφρά οχήματα, χρειαζόμαστε τα super credits, δηλαδή τα οχήματα που εκπέμπουν ε, λίγο. Από όσο γνωρίζω, μια γαλλική βιομηχανία θα ε, κατασκευάσει ηλεκτρικά οχήματα και αυτό είναι πολύ ε, χρήσιμο, δηλαδή να έχουμε κάτω από 50 γραμμάρια και όχι κάτω από 50%. Τα ηλεκτρικά φορτηγά, αν χρησιμοποιηθούν, μαζί με τον, νόμο, τον πράσινο νόμο περί δημοσίων προμηθειών, όλα αυτά θα βοηθήσουν το περιβάλλον. Θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο στόχο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, με τα ποσοστά, να ενισχύσουμε την καινοτομία και αναμένω τις τροπολογίες συμβιβασμού της Επιτροπής σας. Δυστυχώς δεν σας είδα πριν, κυρία Μέρκης, ε, πολύ σύντομα παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους προηγούμενους ομιλητές που μίλησαν για φιλόδοξες ε, προτάσεις. Μιλάμε για την τεχνολογία η οποία είναι έτοιμη όταν είναι ε, έτοιμα και τα πολιτικά μέτρα καθώς και τα μέτρα ρύθμισης. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Μιλώ για 125 γραμμάρια λοιπόν, που είναι κάτι το πιο φιλόδοξο από την Κομισιόν. Και εμείς ε, μιλάμε για όριο ταχύτητας 100 χιλιόμετρα την ώρα. έτσι ώστε να έχουμε 67% απόδοση ως προς την απασχόληση σε δύσκολους καιρούς, πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε νέους τύπους εργασίας, νέο τύπο απασχόλησης. Μιλάμε δηλαδή για μια νέα φιλόδοξη εποχή. Μην αποδυναμώσετε λοιπόν τον κανονισμό όπως ορίστηκε από την Επιτροπή. Νομίζω θα μπορούσε να ήταν και πιο φιλόδοξος θα πρέπει ναι, να καινοτομήσουμε να, και να ρυθμίσουμε με θάρρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσείς κύριε Λάγκεν τώρα σύντομα. Ναι, θα είμαι σύντομο. Εξεπλάγει με την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάνει προτάσεις και μετά έρχεται και ζητεί από το Κοινοβούλιο να είναι πλέον φιλόδοξο από την ίδια. Πολύ παράξενο. Ποτέ δεν μου έχει ξανατύχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ίδια δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υποστηρίζονται τις ίδιες τις προτάσεις. Θα πρέπει να τεθεί το θέμα ποιο εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους που τάσσονται υπέρ μιας κάπως πιο διαφοροποιημένη ερμηνείας. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι, ο κοινός στόχος μας είναι να μειωθούν οι εκπομπές και να ε, υποβάλουμε και στην Κομισιόν και στη βιομηχανία μια πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, λύση με τις απαραίτητες μεταβατικέ περιόδους. Είναι σωστό. Για τα αυτοκίνητα οχήματα, για το διοξίδιο άνθρακος δηλαδή, τα συζητήσαμε με παρόμοιο τρόπο και η ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε τελικά να υπάρξει μια μεταβατική προσαρμογή, το δέχτηκε η βιομηχανία και τελικά είναι μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε παρά να ήμασταν πιο αυστηροί. Τώρα τίθεται το θέμα των super credits και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Να το συζητήσουμε αν είναι καλύτερα 50% ή 50 γραμμάρια. Η δική μου συμβαστική τροπολογία προτείνει 50% που εγώ το θεωρώ ότι είναι καλύτερο διότι δεν μιλούμε για μικρά αυτοκίνητα για, τη μεταφορά προσώπων αλλά για ε, ε, φορτηγά οχήματα μέχρι 3,5 τόνων. Η προώθηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ευκαιρία και επιστώσεις για την ε, κατασκευή μικρών ε, φορτηγών αυτοκινήτων, τότε έχει καλώς. Ναι. Η κυρία Χόλ και ο κύριος Ζαντό ρώτησαν τι γίνεται με τις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτές είναι βέβαια δικές μου τις οποίες έχω πονήσει στην βάση 219 τροπολογιών, οι οποίες μετά από την ε, ε, συνεδρία της Επιτροπής θα σας διαβιβαστούν αμέσως για να μπορέσετε βεβαίως να τις μελετήσετε και να ε, σχηματίσετε άποψη. Η ψηφοφορία προβλέπεται για το τέλος του μηνός και θα υπάρχει χρόνος και για συζητήσεις διμερώς αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο. Η οικολογική δέσμευση της κύρια Φόρντ θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς εάν θεωρούμε ότι δηλαδή οι, περιορι... οι συσκευές περιορισμού ταχύτητας είναι κάτι σημαντικό. Εγώ κύριε Βαν δεν είπα ότι είμαι υπέρ. Ίσως κακώς το κατανοήσατε ή ίσως κακώς σας το μετέφρασαν. Εγώ λοιπόν δεν υπήρξα θετικός υπέρ των συσκευών αυτών, μείωση της ταχύτητας και εν τέλει θεωρώ ότι θα καταλήξει η πλειοψηφία σε εύλογες αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν για το χρονοδιάγραμμα τώρα ακόμη. Η επόμενη συζήτηση γίνεται στις 7 Απριλίου, λέει ο Πρόεδρο. Η πρώτη έγινε 7 Απριλίου βεβαίως, είναι παρελθόν ήδη. 24 Ιουνίου η επόμενη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούλιο. Εδώ λοιπόν λίγη συζήτηση του θέματος αυτού. Θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Ντεκαστήγιο να, αναβάλει, να αναλάβει συγγνώμη, την διεύθυνση συζητήσεως. Please, colleagues. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Καθίστε στις θέσεις σας. Iniciar, eh, la... Αρχίζουμε συναδελφοί τη συζήτησή μας με την Επίτροπο που ασχολείται με την ψηφιακή ατζέντα και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Την κυρία Κρούς θα μας μιλήσει για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης που προετοίμασε η Επίτροπη και θα μας την παρουσιάσει καθώς ε, και του συμβιβασμούς οι οποίοι επήλθαν με βάση δηλαδή και τους συμβασμού οι οποίοι επήλθαν εδώ στη δική μας Επιτροπή. Θα μιλήσουμε για τους μεγαλύτερους ε, στρατηγικούς στόχους και εμβληματικούς της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Um, uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ε, αυτής του Κοινοβουλίου, είναι πραγματικά αληθές ότι σας είχα υποσχεθεί ότι θα ήταν καλύτερο να ειδωθούμε το γλυκορότερο δυνατόν για να σας ενημερώσω το θέμα αυτό. Η πρόταση της ε, ε, Επιτροπής που ξέρετε ευθύθηκε στις 19 Μαΐου είναι το κυριότερο θέμα για την Ευρώπη του 2020. Και αυτό έγινε μόλις ε, τρεις μήνες μετά που έδωσε την υποσχέτη ο κ. Παρόζο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά συμβάλλατε πάρα πολύ σημαντικά κυρίως ε, η κυρία Πιλάντα Καστήριο και οι σκιώδεις συγγητές. Αντίνα Φελέαμ, Κεφάλαιον Κάλβι και Φιλίπ Λομπέαχα. Βλέπετε πολλά που υπάρχουν εδώ στην ε, ε, ψηφιακή ατζέντα, όπως λέμε. Ξέρετε ότι εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, έχουμε παρόμοιες ανησυχίες και οπωσδήποτε είναι σαφές ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Δηλαδή η βελτίωση για τους πολίτες της Ευρώπης. Η ψηφιακή ατζέντα καλέπτει 7 τομείς η αύξηση του κυβερνού εγκλήματος, δίκτυα, έλλειψη διασύνδεση των δικτύων, ευνεπαρκής προσπάθειας κοινοτομίας, έλλειψη των ικανοτήτων για την ε, χρήση των μέτρων αυτών, νέες προκλήσεις και θα ήθελα να συμφωνήσετε να μπούμε για κάθε θέμα στις λεπτομέρειες. Πρώτον, η επίτευξη μιας ζωντανής ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς όπου τα ψηφιακά αγαθά και οι υπηρεσίε θα μπορούν να κυκλοφορούν εξίσου σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά το περιεχόμενο, απλούστευση όσον αφορά το copyright και επίσης τις ε, διασυνοριακές ε, αδειοδοτήσεις για να μπορέσει έτσι να είναι άμεση η επικοινωνία πέρα από τα σύνορα και να υπάρχει όπως έχουμε ένα ενιαίος ε, ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών. ΣΕΒΑ. Εκεί μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, ε, αλληλολειτουργικότητα που είναι το επόμενο σημείο. Λειτουργικότητα και πρότυπα. Υπάρχουν ακόμα πολλές αδυναμίες όσον αφορά τις δημόσιες αγορές, συντονισμό μεταξύ των δημοσίων αρχών και γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερα ICT. Θα θέλαμε να προτείνουμε διάφορα ε, ένομα μέσα για να επιτρέψουμε τα πρότυπα να αναπτυχθούν από παγκόσμιου ε, επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την αλληλολειτουργικότητα προτείνοντας μια στρατηγική για την ευρωπαϊκή αλληλογικότητα ε, και ένα σχετικό πλαίσιο. Το τρίτο σημείο είναι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη. Κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες μας δεν θα ασπαστούν τεχνολογία την οποία δεν εμπιστεύονται. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε όλες τις ε, ε απειλές από το έγκλημα στο κυβερνόχωρο ο, μέχρι την κλοπή ταυτότητας. Εδώ πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ πολιτών και δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Το Σεπτέμβριο η Κομισιόν θα υποβάλει μια πρόταση για εξυγχρονισμένα ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ασφάλεια και την προστασία κατά των κλοπών των ε, συστημάτων πληροφορική και ελπίζουμε ότι όσο συνομοθέτης θα μας βοηθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για την προστασία των ε, δεδομένων. Η Κομισιόν προσπαθεί να προωθήσει την ασφάλεια στον τομέα αυτό της τεχνολογίας με κάθε μέθοδο. Δεν θα περιοριστούμε σε νομοθετικά μέτρα μια ανακοίνωση για την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια θα σας μεταβαστεί αργότερα. Ο επόμενος τομέας αφορά τη γρήγορη και την υπερβολικά γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχει ο στόχος αυτό για το 2015. Και θα πρέπει να εγγυηθούμε ε, γενική πρόσβαση με ταχύτητες μέχρι 30 MB ανά δευτερόλεπτο και σαν ένα απότερο στόχο 100. Η αστική ανακοίνωση που θα υιοθετηθεί κατά διάρκεια του έτους θα παρουσιάσει το κοινό πλαίσιο για να πληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Επίσης, θα προτείνουμε μια φιλόδοξη πρόταση για ένα πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό φάσμα τεχνολογίας με πρωτοτεραιότητα μέχρι το 2015 και καθορισμό συγκεκριμένων ε, μέτρων σε διαβούλευση μαζί σας με τα κράτη-μέλη και με τους ενδιαφερομένους συμπερασμένου και της διάσκεψης κορυφής για το φάσμα αυτό που, θα οργανώθηκε από το Κοινοβούλιο και από εμά από κοινού τον Μάρτιο και μας έδωσε πολλές ιδέες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν προωθεί πιο αποτελεσματική και ευέλικτη χρήση του φάσματος. Και ο συνομοθέτης με τη βοήθεια της Κομισιόν θα μπορέσετε νομίζω να πετύχετε μία λογική συμφωνία πάνω στις πολιτικές προτεραιότητες για 2015 και τους συγκεκριμένους στόχους. Η σύσταση για την πρόσβαση της επόμενης γενιάς θα δώσει ε, κατευθύνσεις στις εθνικές διακανονιστικές αρχές για να ε, εγγυηθεί την πρόσβαση, εξασφαλίζοντας όμως και την ασφάλεια και θα συμφωνείτε μαζί μας φαντάζομαι ότι είναι ουσιαστικότατο εδώ τα συμφέροντα των καταναλωτών. Πέμπτος ε, τομέας είναι η αύξηση της ε, έρευνας και των στην Ευρώπη στον τομέα της πληροφορικής. Ξέρετε ότι η Ευρώπη δεν ε, ε χρηματοδοτεί επαρκώς, κατακαιρματίζει τις προσπάθειές της και έτσι δεν μπορεί να ωφεληθεί από τις προσπάθειες που καταβάλει. Ιδίως αργούμε ε, τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφερθούν σε προϊόντα, να μεταφραστούν σε προϊόντα που θα ωφελήσουν τους καταναλωτές. Και γι' αυτό ε, η Κομισιόν προβλέπει μια σχετική πρωτοβουλία, της οποίας ε, ηγείται ο συνάδελφος Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά έχουμε συγκεκριμένους στόχους για την πληροφορική θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις και να συνεργαστούμε καλύτερα με τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να διπλασιάσουμε το ετήσ, τις ετήσιες δαπάνες μέχρι 11 δις ευρώ για το 2020 στον τομέα της έρευνας. Προτείνουμε επίσης μεθόδους για πιο εύκολη και γλύχωρη πρόσβαση των ΜΜΕ και νέων ευρωντικών ερευνητών συγγνώμη, στους πόρους αυτούς έρευνας. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε το να γνωρίζουν όλοι τα θέματα της πληροφορικής, γιατί ξέρουμε ότι η έλλειψη αυτής της ικανότητας εξακολουθεί να παρεμποδίζει την ανάπτυξη της οικονομίας. Παρόλα την πρόοδο, το 30% των Ευρωπαίων δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. παρθένες της πληροφορικής, αν μπορώ να το πω έτσι. Και έχουμε μεγάλη έλλειψη για την κάλυψη των θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτό που θα φτάσουμε μέχρι 700.000. Άρα χρειαζόμαστε καλύτερα να εστιάσουμε τους πόρους της Ένωσης και αυτό θέλουμε να το κάνουμε με το να συμπεριλάβουμε τις ικανότητες αυτές της ε, χρήσης ε, της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών προγραμμάτων. Αλλιώς δεν θα ωφεληθεί η ευρωπαϊκή κοινωνία από την πρόοδο στην πληροφορική. Έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση παραδείγματος χάρη της κλιματολογικής αλλαγής ή της γέρασης του πληθυσμού κλπ. Η πληροφορική για το περιβάλλον, Φελιππίν. Η πληροφορική θα μπορεί να είναι ένα σημαντικό εταίρο για την βελτίωση τη αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να δούμε πώς έχουν υιοθετηθεί όλα αυτά και πώς θα προωθήσουμε την διαλειτουργικότητα. Η κύρια πρόκληση είναι να έχουμε δημόσιες υπηρεσίες online που θα λειτουργούν ε, διασυνοριακά. Και επίσης θα αναπτύξουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης για το 2010 για να αναφέρεται στους κύριους στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια για την κινητικότητα στην εσωτερική αγορά. Όταν αναφερόμαστε στη γύρωση του πληθυσμού και στις ε, τεχνολογίες πληροφορικής, αναφερόμαστε σε εκείνους που χρειάζονται ενίσχυση στην καθημερινή του ζωή. Ένα πρόγραμμα που αρχίσαμε πριν από δύο χρόνια με έντονη υποστήριξη από εσά και που φαίνεται ότι προχωράει πολύ καλά. Εγώ ξεκίνησα μια προσωρινή αξιολόγηση του προγράμματος για να δούμε πώς έχει προχωρήσει και θα σας κάνουμε μια παρουσίαση και σας και το Συμβούλιο προφανώ μέχρι τα τέλη του έτους. Σίγουρα θα σημειώσατε ότι πολλά από τους τομείς αυτούς που ανέφερα εδώ έχουν σημαντικές διεθνείς επιπτώσεις. Γιατί πολλά από αυτά μπορούν να προωθηθούν μόνο σε διεθνές επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καλή διακυβέρνηση του διαδικτύου όσο καλύτερα μπορούμε να συνεχίσουμε το διακυβερνικό φόρουμ που είναι σημαντικό στο τομέα αυτό και χαίρομαι που ο Φρανσίσκο Σούζα Βάγνερ το περιλαμβάνει στην έκθεση που θα παρουσιάσει. Ελπίζω σε επόμενες εβδομάδες να βρείτε τους συμμετέχοντες στην επόμενη διασκέψη στο Φούλνες το Σεπτέμβρη για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να κάνουμε ό,τι πρέπει ούτως ώστε η, η διάσκεψη αυτή στο φούρνο να είναι επιτυχής. Πρόκειται για ένα πολύ πολύπλοκο και φιλόδοξο πρόγραμμα και ε, χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα προηγουμένως, πράγμα που προϋποθέτει καλή και φιλόδοξη εφαρμογή των δομών. Ξέρω ότι θα είστε πολύ επικριτικοί για την δομή αυτή. Ο πρόεδρος της Κομισιόν όρισε μία ομάδα ε, επιτρόπων για τη ε, ψηφιακή αυτή τεχνολογία για να μπορέσει να εξασφαλιστεί με τη βοήθεια των κρατών μελών οι προσπάθειές μας να καταπτύσσονται επαρκώς σε εθνικό επίπεδο και επίσης και από εσά εδώ στο Κοινοβούλιο και από όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα μπορούμε να δούμε την πρόεδρο στην, ε, στην ε, ατζέντα μας αυτή με ετήσιες αξιολογήσεις και συνενώντας όλα τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους θεσμούς και, και ενδιαφερόμενους για να συζητήσουμε το αποτέλεσμα. Και τέλος, σε συμφωνία με την, ε, τους στόχους του 2020, του 2020, θα σας κάνουμε ετησίως μια παρουσίαση και ιδίως και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προσβλέπω στη συνεργασία σας για να πετύχουμε αυτό το τόσο φιλόδοξο ψηφιακό χρονοδιάγραμμα Ορισμένα συμπληρωματικά σημεία για το πρόγραμμα εργασία. Ξέρω ότι είναι κάπως ρηψοκίνδυνα όλα αυτά που προτείνουμε. Αλλά θα ήθελα να συζητήσω κάποια από τα θέματα αυτά όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος για, την, για τον τηλεοαναγωνισμό. Σύντομα θα σας παρουσιάσω μία προσωρινή ε, έκθεση όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ξέρετε ότι ο δεύτερος σχετικός κανονισμός γλίγορα επιβλήθηκε και υπάρχουν χαμηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή για τη τηλεφωνία παρόλα αυτά απαιτούνται περισσότεροι πρόοδοι. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου. Είχα πει ότι θα έχουμε νέους χρήσιμους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να αποφύγουμε να δίνουμε βεβαιασμένες απαντήσεις πριν έχουμε αξιολογήσει πλήρως τα προβλήματα και κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα γιατί θα πρέπει να μιλούμε για τον ίδιο ορισμό της ουδετερότητας του δικτύου. Αλλιώς θα δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα από εκείνα που προσπαθούμε να λύσουμε. Προς το στόχο αυτό θα ξεκινήσουμε μια ε, δημόσια διαβούλευση πριν από τις θερινές διακοπές για να δούμε κατά πόσον άλλες συμπληρωματικές ε, διακανονιστικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες ή όχι. Πάντως, οπωσδήποτε, οι κατευθυντήριε γραμμέ που θα ακολουθήσω είναι καταρχήν ελευθερία έκφραση, ουσιαστικότατη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Διαφάνεια, δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τρίτον, χρειαζόμαστε ε, επενδύσει σε αποτελεσματικά και ανοιχτά δίκτυα και τέταρτον, δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε ε, ορισμένες πρακτικές που έχουν σαν στόχο τον, την παρεμπόθεση του ανταγωνισμού και τέλος θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ε, αποτελεσματικά συστήματα επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίε μας ασχολούνται και με τον διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα αυτό. Το είχαμε πει και νωρίτερα φέτος την Άνοιξη. Ξέρετε ότι γίνεται αυτές οι διαπραγματεύσεις για τη δέσμη Telecom μετά από εκείνα που είχαμε το 2009. θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι διατάξει της Ευρωπαϊκής για τις ε, ε, σφαιρικές υπηρεσίες έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ανάπτυξη για όλους. Οι ανοιχτέ διαβουλεύσει που άρχισαν στις 7 Μαου είναι τώρα διαθέσιμα τα αποτελέσματά τους στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με την ανάλυση των συμβολών και θα ήθελα να είμαι σαφής, τονίζοντας ότι δεν έχω καμία προκαταρκτική δυνατότητα προσαρμοσμού αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξεταστεί σε έναν ασαφή ε, χώρο χωρίς να σχετιθεί με τα κοινωνικά, οικονομικά και άλλα θέματα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι όλα λέβετα. Θα πρέπει να τα εκτάσουμε στο σύνολό τους. Και αυτό ισχύει για το σύνολο της ε, ψηφιακής ατζέντα. Όλα είναι αλληλένδετα και με τα κοινωνικά θέματα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξεταστούν μετά από τα αποτελέσματα της δέσμης Telecom του 2009 με την προοπτική του 2020 και με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Το φθινόπωρο θα υπάρχει μία έκθεση όσον αφορά τελικά αποτελέσματα της διαβούλευσης και εάν χρειαστεί να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις για την βελτίωση της οδηγίας για τις σφαιρικές και νοφιλές υπηρεσίες, θα το εξάσουμε τότε. Αυτή τη στιγμή είναι πρόωρο να κάνουμε οτιδήποτε. Σήμερα το πρωί είχαμε μια δια... ένα συμβούλιο τηλεπικοινωνίας και αν μου επιτρέπετε να σας προσθέσω κάτι για τα αποτελέσματα, έχω να σας πω ότι οι Υπουργοί υιοθετήσαν τα συμπεράσματα για την ε, ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη και ε, υποστηρίζουν τώρα τις κύριες ε, δράσεις προτεραιότητας που αναφέρονται στην πρότασή μας. Επίσης, σαν προς τα κράτα-μέλη και τις κυβερνήσεις τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα λάβουν υπόψη επίσης μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το 2020. Θα ρίνουν λοιπόν τον ε, οριζόντιο συντονισμό και σε κοινοτικό και σε ε, εθνικό επίπεδο για να βελτιωθεί η εφαρμογή της ατζέντα αυτής και παρόλο που είναι θαυμάσιο που υποστήριξαν την ψηφιακή αυτή ατζέντα, είχα την ιδιαίτερη δυνατότητα ούτως ώστε να τους κινητοποιήσω γιατί ξέρω ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε εσείς και εγώ χωρίς τους υπουργούς, χωρίς τα κράτη-μέλη. Πρέπει εκείνοι να εφαρμόσουν αυτά που αποφασίσαμε σήμερα. Πρέπει να τα εφαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι λογικός και να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Επίσης, είχαμε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψη για το πώς καλύτερα θα δώσουμε στους πολίτες Ευρώπης απλή και εύκολη πληροφόρηση όσον αφορά τα δικαιώματά τους μέσα στα πλαίσια της ε, ε, πληροφορικής. Δηλαδή να αυξηθεί έτσι η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών στο διαδίκτυο. Τι, όπως σας είπα και προηγουμένως, εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε έτσι να ενθαρρύνουμε τους πάντες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Παραδείγματο χάρη, τράπεζε, online αγορές κλπ. Χρειάζεται όμως για όλα αυτά εμπιστοσύνη. Στο Συμβούλιο σήμερα καθορίστηκε στη Ρήγα η έδρα της υπηρεσίας αυτής που τη χαίρομαι γιατί η κυβέρνηση της Λετωνίας έκανε μια ωραία προσφορά θα έλεγα όχι μόνο για την τοποθεσία αλλά μας προσφέραν ωραία γραφεία και υλικό και λογισμικό μας δίνουν λοιπόν πολλά για να μπορέσουν έτσι να συμβάλλουν σε ένα καρποφόρο μέλλον γιατί η ώρα συνεδρίαζε στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση της Λετωνίας όμως είπε ότι θα αναλάβουν και τα γραφεία αυτά τα συμπληρωματικά που χρειάζονται για να μπορέσουν να λαμβάνουν χώρα εκεί αυτές οι συνεδριάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι η τελευταία αναλύση είναι καλό αυτό και ευχαριστώ τις αρχές της Λετωνίας για την προσφορά τους. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ε, Επιτροπή Διαχείρισης του ΠΕΡΑΚ έκανε τη δεύτερη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα και επέλεξαν κάποιους υποψηφίους. Πρόκειται για τον Αντορέμα, έναν εστονό, ο οποίος θα έρθει αν τον καλέσετε για να σας, σας και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την εμπειρία του μέχρι στιγμής και για το τι θα πρέπει να γίνει. Το Μπέρεκ λοιπόν είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις εργασίες του και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και πολλά πρέπει να γίνουν και θα θέλετε φαντάζομαι με όλα αυτά τα σχέδια για το 2007, ε, 10 συγγνώμη, και όποτε θέλετε να μου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Και είναι σαφές θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα μέσα για την εφαρμογή αυτών που όχι μόνο ελπίζουμε, αλλά που εξηγούμε προς τους Ευρωπαίους πολίτες που, ότι πρέπει να γίνει για να νομίζουμε την κρίση. Η ψηφιακή ατζέντα λοιπόν είναι μια καλή εναλλακτική για υγιές μέλλον. Τούτου λεχθέντος, αυτά που έκανα σήμερα είναι ότι έδωσα αυτές τις πλαστικές κάρτες σε όλους τους υπουργούς. Ε, είναι λίγο κίνδυνος αυτός βέβαια, γιατί αυτή είναι μια κάρτα που σε δύο, σε δύο γράφει ακριβώς τι πιστεύουμε και τι θα κάνουμε. Μπορείτε να το πάρετε λοιπόν, είναι πραστικοποιημένο, δεν μπορείτε να το σκίσετε, να το καταστρέψετε και θα σας δώσω τις κάρτες αυτές και για σας, σε εσά. Αν δεν είναι αρκετές θα σας δώσω και άλλες άμα θέλετε να μου τις ζητήσετε απλώς. Ε, κυρία Αγαπητέ Αγαπητοί Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμέναμε αυτό το έγγραφο, αυτή την ανακοίνωση εδώ και πολύ καιρό και μας το παρουσιάσατε στην Επιτροπή, στην Ήτρε, στην Επιτροπή μας με μεγάλη θέρμη και κάθε φορά ε, είσαστε ευπρόσδεκτοι γνωρίζετε τη θέση σας σε αυτό το θεσμικό όργανο που είναι μέρος του οίκου σας, θα μπορούσα να πω, ιδιαίτερα η Επιτροπή μας, η Ήτρε. Έχουμε έναν ε, κατάλογο συναδέλφων, ένα μακρύ κατάλογο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο κλείνουν. 16, 16. Ε, αν υπάρχει κάποιος άλλος να μου το πει τώρα. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε πόσοι θα παρέμβουν, πόσοι είναι οι ομιλητές. Με την κυρία Φόρντ 16 είναι οι ομιλητές. Κλείνει ο κατάλογος. Θα έχουμε τρεις γύρους για να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα για την Επίτροπο, για τις απαντήσεις 5, 5 και 6 Αρχίζει ο πρώτος γύρος και θα ήθελα εγώ να παρέμβω όχι ως ε, πρόεδρος, ε, προεδρεύουσα αυτής της συνεδρίασης, αλλά ως βουλευτή σε θέματα ψηφιακής ατζέντα, επειδή θα ασχοληθώ και εγώ ως εισηγήτρια με το θέμα. Εντάχει λοιπόν, νομίζω ότι με την πρόταση αυτή της Κομισιόν βλέπουμε πώς έχει αυτή η αποστολή, πώς προσδιορίζεται για να φτάσουμε σε μία πλήρη ψηφιακή ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει θέμα συνεργασίας βεβαίως με τη δική μας έγκριση του πλαισίου στις 5 Μαΐου και με τις προτάσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου υπό Ισπανική Προεδρία τώρα και πριν υπό Σουηδική που ήταν ιδιαίτερα δραστήρια σε αυτό το τομέα. Κάτι το οποίο είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο. Τώρα ήρθε η ώρα να δράσουμε έληξαν οι συζητήσεις για το περιεχόμενο της ψηφιακής ατζέντα και φτάνουμε στη δράση για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτή την ψηφιακή ατζέντα, να την πραγματώσουμε. Υπάρχουν πολλές ε, υποδείξεις προς την Επίτροπο που είναι σημαντικές και αναφέρθηκαν, έχουν προαναφερθεί. Θα ήθελα όμως καταρχήν να τονίσω την ανάγκη μίας τάχης της μεταφοράς του πακέτου Telecom. Γιατί είναι πρόκριμα, αποτελεί πρόκριμα για την ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντα και χωρίς ε, αυτή την προϋπόθεση η ψηφιακή ατζέντα θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και ελλείψεις. Δεύτερον, από πλευράς ε, καθαρά προτάσεων από, πλευράς, από την πλευρά της Κομισιόν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη θέματα χρονισμού με την ατζέντα. Όπως μας είπε και η Επίτροπος, χωρίς ε, περαιτέρω καθυστερήσεις, διότι εδώ και ένα χρόνο πια, κλείνουμε ένα χρόνο θητείας Δυστυχώς καθυστέρησε η ανάληψη καθηκόντων για τους γλώσσους που γνωρίζετε. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε. Ό,τι εξαρτάται λοιπόν από το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής ατζέντα στα πλαίσια της ευρυζωνικότητας ε, τελεκόμ ή ουδετερότητας των δικτύων, δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε καθόλου από τη στιγμή θέση σε ισχύ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω εν μέρει και το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων. Σε σχέση με την ουδετερότητα του δικτύου, η ίδια η ατζέντα της Κομισιόν κάνει λόγο για την ανάγκη επιμερισμού, συγχρηματοδότησης, όπως ισχύει και με τις τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε για γεωγραφικό ε, διαχωρισμό ή κατακαιρματισμό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν όλες αυτές τις αρχές που ίσχυσαν και στο πακέτο Telecom. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο ζωτικής σημασίας για να αναπτυχθεί η ψηφιακή ατζέντα χρειάζεται όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά και η συμμετοχή άλλων γενικών διευθύνσεων, άλλων χαρτοφυλακίων, άλλων επιτρόπων. Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ψηφιακή ε, ενιαία ατζέντα ως ανοιχτή ατζέντα. Άλλες επίσης ελευθερίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και η ΙΝΚΟ θα πρέπει να ασχοληθεί δηλαδή με την ε, προστασία των καταναλωτών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλυφθούν εγκαίρως, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως. Γι' αυτό η Επίτροπος έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να κατέχετε ηγετική θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να δράσει άμεσα η Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή υπό την αιγίδα σας στην Κομισιόν να προωθηθεί αυτό το θέμα, μέσα και από άλλα χαρτοφυλάκια έχω, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γνωρίζω ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε, μπορείτε να βασιστείτε και σε εμά προς αυτή την κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλες στη συνέχεια. Στην παρέμβασή σας, κυρία Επίτροπε, είπατε ότι το θέμα της ασφάλειας είναι από τα κρίσιμα θέματα της ψηφιακής ατζέντα. Έχω μία ερώτηση σχετικά με την οργάνωση εργασίας της Κομισιόν. Θα υποβάλλεται φέτος έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Ίντερνετ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δεν έχει καν δική της ε, σύνδεση με το ίντερνετ και δεν παίζει κανένα ρόλο για την ώρα παγκοσμίω. Υπάρχουν και Αμερικανοί οι οποίοι Αμερικανοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος προβλέπει επένδυση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ασφάλεια του ίντερνετ. Για φέτος προβλέπουν 300 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το Security Act προβλέπει επίσης και την προτροπή προς το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρώπη για να συζητήσει κοινά πρότυπα ασφάλειας. Εμείς χρειαζόμαστε λοιπόν ρυθμίσεις και εδώ στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε ισότιμα με τους Αμερικανούς για την λεγόμενη κυβερνοασφάλεια. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν και πάλι στον σχεδιασμό του νόμου της ΙΝΙΣΑ, δηλαδή της, του οργανισμού μάλλον ασφάλειας του ίντερνετ, να προβλέψετε τα σχετικά, διότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ισοδύναμοι με τους Αμερικανούς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει ε, να υπαχθούν σε μια ενιαία σε ένα νέο σχέδιο, ένα ενιαίο κόνσεπτ. Γιατί και εδώ θα προερθούν 30, 40, 50 εκατομμύρια για την ασφάλεια του ίντερνετ, του διαδικτύου και για τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Βιομηχανία θα παίξει ένα ρόλο η ε, ασφάλεια του διαδικτύου. Εκτός λοιπόν από την δική σας ψηφιακή ατζέντα και το θέμα ασφάλειας, θα ζητήσω να υπάρξει και μια ανακοίνωση ή πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη ενός κόνσεπτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα συνεργαστούν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις και ποιο θεσμικό ρόλο θα παίξει στο μέλλον ο Οργανισμός Ασφάλειας του Διαδικτύου. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, λέει κυρία Τράουτμαν, που προσήλθατε εδώ για να μας μιλήσετε για την ψηφιακή ατζέντα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Υπάρχει θέμα διαλειτουργικότητας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά ως προς τα ανοιχτά πρότυπα είδα ότι σε μία ενδιάμεση έκδοση η ανακοίνωση μιλά για το ελεύθερο λογισμικό ως ε, ε, βασικό στοιχείο για την μελλοντική ψηφιακή ατζέντα και δεν βλέπω τις ίδιες διευκρινήσεις τώρα, δηλαδή δεν γίνεται πια μνήα στο ελεύθερο λογισμικό. Και πάλι ως προς αυτό το σημείο, γιατί έχει επέλθει αυτή η αλλαγή σε σχέση με την ενδιάμεση διατύπωση και την τελευταία. Ως προς τις διατυπώσεις που αφορούν την τεχνολογία, δηλαδή τις, ραδιοσυχνε... τις ραδιοσυχνότητες. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το ουδέτερο πλαίσιο να μην το έχουμε ως ε, ε, μία ανοιχτή πόρτα προς τις μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες και να δώσουμε μία ευκαιρία και στις δικές μας τεχνολογίες που είναι ε, καρπός των δικών μας προσπαθειών στον τομέα του R&D, του ελεύθερου λογισμικού και των ουδέτερων δικτύων. Θα πρέπει να βρει μία διέξοδο σε σχέση με τις βιομηχανικές διεξόδους των καινοτομιών μας, η ψηφιακή ατζέντα είναι περίπλοκη, αλλά ως προς τα δίκτυα αυτά ε, θεωρείτε ότι έχουμε χάσει εκ των προτέρων ή βασίζομαστε σε μία ενδυνάμωση του ηγετικού μας ρόλου σε σχέση ε, με τους παρόχους και την απόδοσή μας ως προς τις online υπηρεσίες, δηλαδή το, το τρίτο αυτό στρώμα. Έχω και άλλες ε, δύο ερωτήσεις. Η κυρία Πιλάρντε Καστίγιο αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Ποια είναι τα μέσα που διαθέτει η Επίτροπη για τη μεταφορά του πακέτου Telecom. Ξέρω ότι έχετε πολύ καλές προθέσεις, αλλά ποια μέσα θα ε, προωθήσει η Κομισιόν προς αυτή τη μεταφορά, διότι ορισμένα κράτη-μέλη μεταφέρουν ε, παίρνοντας και ορισμένες ε, ελευθερίες. Πέρσι μας ανακοινώσατε ένα πλαίσιο μέτρων Εάν δούμε τη διαδικασία διαβούλευσης βλέπουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις παλινδρομούν σε σχέση με τις επενδύσεις ε, που είχαν προκριθεί. Μπορείτε να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πώς, πότε θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση και σε αυτή την ε, χρηματοοικονομική κρίση. Και αυτό αφορά και την ευρυζωνικότητα, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει μια νέα όθηση. Ο κύριος Βούι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στο άρθρο 2 της Digital Agenda λέτε θα πρέπει ε, να μέσα στα εθνικά και διεθνή τέλη περιαγωγής να υπάρξει μηδενικό στόχος μέχρι το 2015. 2015 βέβαια είναι ακόμα αρκετά μακριά, δηλαδή είναι 4-5 χρόνια ακόμη μέχρι ό,τι επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Από την άλλη μεριά βρισκόμαστε τώρα στις δημοπρατήσεις ε, των ευρέων φασμάτων και είπατε ότι θα φτάσουμε και μέχρι 100 MB το δευτερόλεπτο. Το 1 MB μέχρι τώρα είναι λιγότερο από ένα λεπτό του ευρώ. Από την άλλη μεριά για την ίδια ε, για την ίδια σε προσφορές υπηρεσιών χρεώνονται μέχρι και 19 λεπτά. Τώρα, Θα μειωθούν επίσης τα 80 ε, λεπτά για την ίδια περίοδο. Επομένως για τα 100 ΜΒ το δευτερόλεπτο, αν πάρουμε τα 19 ευρώ, φτάνουμε στο ένα δευτερόλεπτο για 1900 ευρώ. Φτάνουμε στα 1900 ευρώ για ένα δευτερόλεπτο. Τι θα πούν τότε οι πολίτες μας για αυτές τις προσφορές υπηρεσιών. Εμένα με ενδιαφέρει, βεβαίως υπάρχει μια τεράστια αύξηση του όγκου δεδομένων και κυρίως στα μηχανήματα τέταρτης τεχνολογίας, αλλά και για τα ε, δίκτυα των 800 MHz, αλλά ποια βήματα προτείνετε για το μέλλον. Και νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να κινηθείτε πάρα πολύ γρήγορα. Το δεύτερο σχόλιο μου, και εδώ σας επενώ επίσης, για το ότι προτίθεστε να κάνετε διπλασιασμό των επενδύσεων του δημόσιου τομέα, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι δημοπρατήσεις που γίνονται για την ώρα δίνουν ε, κίνητρα για τις χώρες μέλη εάν επενδύσουν και πάλι δηλαδή τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις αυτές πάλι στο, ε, στον ίδιο τομέα, δηλαδή για παράδειγμα με κοινοπραξίες στη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή να δοθούν άλλα κίνητρα, ούτως ώστε ο όγκος των επενδύσεων να αναπτύσσεται διαρκώς. Ευχαριστώ Παουλ. Τελευταίος σε αυτό τον γύρο, ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, ο πρόεδρος Μπαρόσο θα έπρεπε να σας είχε αναθέσει μάλλον την έκθεση για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Γιατί συγκρίνοντας αυτά που έχετε γράψει εσείς με αυτά που έχει γράψει ο κύριος Μόντι, βρίσκω ότι είναι πολύ πιο φιλόδοξα τα δικά σας. Και εσείς εγκρίνατε, ακόμα και για την Digital Agenda μόνο, μια ευρεία προσέγγιση. Αυτό είναι το πρώτο μου θετικό σχόλιο. Ότι εξετάζετε την ICT όχι μόνο ως τεχνολογία καθεαυτή, αλλά ως ένα μέσο για να επιτευχθούν λύσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό για να ξαναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοπόρα θέση της τεχνολογίας. Δεύτερο, όπως είπε η κυρία Τροθμάν, η διαλειτουργικότητα και τα κοινά πρότυπα. Το ελεύθερη πηγής ε, λογισμικό έχει εξαφανιστεί βέβαια από το τελευταίο σας έγγραφο, αλλά το γεγονό ότι εξακολουθούμε να στοχεύουμε σε ανοιχτά πρότυπα, αυτό έχει κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς. Εν τέλει το γεγονός ότι εσείς καθορίζετε ε, συγκεκριμένες προθεσμίες είναι, είναι σωστό δεν σας αρκεί δηλαδή μονάχα να κάνετε σκέψεις. Τώρα, αυτά είναι τα τρία θετικά σχόλια. Τώρα, τρία σχόλια που θα ήθελα να κάνω, που ε, είναι μάλλον το μίσο που με ανησυχούν. Πρώτον, ότι υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός στόχων και είναι δύσκολο να τους παρακαλουθεί κανείς όλους. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μην χάσετε τον προσανατολισμό σας από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν θέλουμε βεβαίως να ξανασυναντηθούμε σε λίγα χρόνια και να διαπιστώσουμε ότι ελάχιστοι από τους στόχους αυτούς επιτεύχθηκαν. Δεύτερο, κάτι που είπε η Πιλάρ σχετικά με την ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή και άλλοι επίτροποι, γιατί πολλούς από τους στόχους που έχετε θέσει εμπίπτουν και στα πεδία αρμοδιότητας άλλων επιτρόπων. Εδώ ανησυχώ κάπως, διότι ενδεχομένως ο Επίτροπος Ποτόσνικ ή η Επίτροπος Έντεγκαρτ ή άλλοι μπορεί να μην είναι απόλυτα μέρος του, της ομάδας πυρήνα της Digital Agenda. Γιατί οι τελευταίοι δύο που ανέφερα ε, είναι πιο πολύ απολύπτες των δικών σας προσπαθειών και θέλετε βεβαίως να συμμετέχουν. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί τη συνάδελφοι, που είναι βέβαια ευκαιρία, είναι όμως και απειλή. Γνωρίζουμε ότι πριν μας πλήξει η κρίση, ήδη είχαμε λίγους ανθρώπους που είχαν τα απαραίτητα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για να ασχοληθούν με την ICT. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο, από 3 μέχρι 700.000 παραπάνω. Υπάρχουν λοιπόν οι ευκαιρίες. Βρισκόμαστε μάλιστα τώρα σε κρίση. Χρειάζεται, χρειαζόμαστε λοιπόν αυτούς τους επαγγελματίες. Και βεβαίω υπάρχουν και λεφτά στον τομέα αυτό όμως είναι και απειλή με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να τους βρει. Αυτούς δεν κρέμονται από τα δέντρα για να πάει να τους κόψει σαν φρούτα. Επίσης τέλος δεν θα πρέπει να ε, εφησυχάζουμε. Εάν δείτε τι είδους ποσά 88 δις από την αμερικανική πλευρά, 37 δις από την ευρωπαϊκή ε, πλευρά Αν δείτε ότι από τις 10 ε, ε, top επιχειρήσεις στον κόσμο, ε, στον τομέα αυτό, μία μόνο είναι ευρωπαϊκή. Εμείς χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, έτσι δεν θα είμαστε επιτυχείς. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, έχετε επιτύχει πολλά μέσα σε ένα τρίμηνο. Σας συγχαίρω για το λόγο αυτό. Βέβαια, θα έχετε την υποστήριξή μας ασφαλώς θα παρακολουθούν προσεκτικά το τι κάνετε, αλλά νομίζω ότι βασικά κινείστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εσείς κυρία Επιτροπή τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα επικοδομητικά και σχόλια επίκριση θα μπορούσα να πω, ή κρίσιμα σχόλια. Γνωρίζω ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ένα οριζόντιο χαρτοφυλάκιο και έχω να κάνω με 26 συναδέλφους. Μιλώντας για τον πρόεδρο πάντα λέω ότι και εγώ τον χρειάζομαι και εκείνος με χρειάζεται. But the other 25, so to say... Αλλά ως προς τους άλλους 25 Όλοι θα πρέπει να εμπλακούν στη συζήτηση, έτσι ώστε να πρόκειται για συνολικό κέρδος. Είμαι αρκετά μεγάλη για να ε, βασίζομαι, ε, να κάθομαι στις δάφνες μου. Το αφήνω για την άλλη μου ζωή. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι οι στόχοι θα εκπληρωθούν δεν λέμε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ούτε είναι ένα από αυτά τα θέματα που θα γίνουν τώρα ή ποτέ ή δεν θα γίνουν ποτέ. Αυτό μας ενέπνευσε μέσα στην ομάδα μου πώς χρόνια μπορούμε να φτάσουμε σε κάτι που είναι σαφές, ε, διακατέχεται από διαφάνεια. Δεν είμαστε ονειροπόλοι Άρα συμφωνώ με όλους σας, ξεκινώντας με την ε, Προεδρεύουσα, την κυρία Ντελκαστήγιο, συμφωνώ ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο το ταχύτερο δυνατόν. Και δεν αρχίζουμε εκ του μηδενός. Είχαμε τη συζήτηση για το πακέτο Telecom που ήταν και το σημείο εκκίνησης και μετά αναλάβατε μια έκθεση για την πολιτική φάσματος και άλλες ειδικέ εκθέσεις. Ξέρουμε δηλαδή στο μεταξύ τι πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το διακύβευμα. Και αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, δηλαδή το ότι θα πρέπει να επιτευχθεί βραχυχρόνια. Αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί εξ αρχής είναι αυτό που συζητήθηκε με τους συναδέλφους και όλοι τα κατάφεραν πολύ καλά. Και αν κατάφερα εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους, αυτό σημαίνει πολλά. Γιατί αναγνωρίζω ότι μέχρι τώρα ήμασταν αποτελεσματικοί. Θα ήθελα να εφαρμόσω ε, μία ψηφιακή ατζέντα επικοινωνιών το ταχύτερο δυνατόν και θα αρχίσουμε με τον πίνακα επιδόσεων και αυτό που έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει με το βαθμολόγιο αυτό. Θα ξεκινήσουμε από εκεί έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα εγκαταλείψει το παιχνίδι. θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί ως προς την κρίση μας. Η κυρία Ντελ Καστήλιο στάθηκε σε αυτό το θέμα που είπατε και εσείς. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τον ουδέτερο χαρακτήρα του διαδικτύου στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. γνωρίζετε εδώ και πέντε χρόνια, ξέρετε ότι πάντα προήγα τη διαφάνεια και τον ουδέτερο χαρακτήρα του διαδικτύου. Άρα ε, έγινε, θα γίνει δημόσια διαβούλευση για το θέμα της ουδετερότητας. Η Κομισιόν θα ζητήσει τη δική σας γνώμη και το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο κύριος Έιλερ μίλησε, διέκοψε η ε, αντιπρόεδρος. Ε, ναι, έφυγε, αλλά θα του τα πείτε εσείς μίλησε για ένα εκπληκτικό ζήτημα. Εκπληκτικό δεν είναι η σωστή λέξη, είναι ύψη της σημασίας, δηλαδή τα θέματα ασφάλειας. Εάν μιλάμε για δίκτυα και ασφάλεια, μιλάμε για επιμερισμένη αρμοδιότητα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, μιλάμε και με τις ΗΠΑ, αλλά μετά το 2006 όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συζητούν για να φτάσουμε σε μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας και γνωρίζουμε ότι είναι ε, ζήτημα επαφών. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας ε, βασίζεται σε μια συνεργατική πολιτική, στην ε, δηλαδή εταιρικότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το ότι δηλαδή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εσείς είσαστε έτοιμοι ως προς την ψηφιακή ε, ατζέντα. Εμείς θα προφάλουμε ορισμένα επιμέρους ζητήματα και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι από κοινού θα τα καταφέρουμε. Γνωρίζω τις στενοπούς, γνωρίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, βασικές ελευθερίες και την ακαιρεότητα και αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε με την ε, ε, ασφάλεια στην Ευρώπη. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας και να φτάσουμε σε μια κοινή πολιτική. Και οι δύο πτυχές αποτελούν ε, ουσία και είναι υποχρεωτική και οι δύο για να καταπολεμήσουμε την απάτη και να ε, προβάλλουμε την τήρηση του νόμου. Η κυρία Τράουτμαν και ο κύριος Λαμπέρ με ρώτησαν γιατί δεν προωθούμε τις ανοιχτές προδιαγραφές, open standards και κατανοώ τι εννοείται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν θα ήθελα να δώσω μάχη ως προς την ορολογία, αλλά ως προς τη δράση. Και αν συμφωνήσουμε ότι η δράση και τα αποτελέσματα αυτής είναι και το πιο σημαντικό, τότε θα προβάλλουμε καλύτερες προδιαγραφές, διότι αποτελούν ένα μέσο προς ένα συγκεκριμένο στόχο και αυτό αφορά και τις τηλεπικοινωνίες και τις πληροφορίες και την διαλειτουργικότητα της ψηφιακής ατζέντα. Ξέρετε από την προηγούμενή μου θητεία τι έκανα στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Για μένα είναι κάτι το απαιτητό και αν λάβουμε υπόψη τις ε, κοινοπραξίες διαδικτύου, οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Δυστυχώς όμως γίνονται ε, διακρίσεις ως προς τις δημόσιες προμήθειες και αυτό κατά της διαλειτουργικότητας. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Είναι απόλυτα σαφές. Θα θέλαμε οι προδιαγραφές να είναι πιο διαφανείς. και επ' αυτού εστιάζουμε την προσοχή μας. Σύμφωνα με την βιομηχανική πολιτική. Η κυρία Τράουτμαντ πολύ σωστά το είπε. Θα αναλάβω δράση εάν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο. Γιατί αν δεχτούμε μία παρόμοια στάση, τότε έχουμε χάσει σίγουρα. σε σχέση με θέματα προσβασιμότητας. Θα προβάλλω διαφανείς προτάσεις το φθινόπωρο. Ορισμένοι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να τύχουν ρύθμισης, αλλά χαμηλής ε, ρύθμισης. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ρύθμισης για τη ρύθμιση, μόνο αν έχει λόγο ύπαρξης και δεν θα θέλαμε να ευεργετήσουμε ε, ορισμένους εμπλεκόμενους ε, φορείς της αγοράς. Εγώ θέλω να ενθαρρύνω ε, τις επενδύσεις για οποιοδήποτε επενδυτή. Δεν μιλάμε για τους υπάρχοντες σε σχέση με τους μελλοντικούς παρόχους. Θέλουμε σαφείς λύσεις έτσι ώστε όλοι να μπορούν να παρεμβούν για να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό. Τους αγαπώ όλους λοιπόν και δεν τάσομαι υπέρ κάποιου συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση δηλαδή. Σε σχέση τώρα με τους ε, στόχους περιαγωγής, οι διαφορές από τους εθνικούς παρόχους και το roaming είναι κάτι που μας απασχόλησε και στο, και στο παρελθόν. Είδαμε ότι δεν υπάρχει πραγματική εσωτερική αγορά στις τηλεπικοινωνίες, το γνωρίζουμε. Άρα αφού το γνωρίζουμε θα βρούμε και μία λύση και τη στιγμή που το κόστος ε, του roaming δεν θα πρέπει να ε, απέχει πολύ από το κόστος των εθνικών παρόχων, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι καταναλωτές υψηλότερες τιμές για την περιαγωγή. Συμφωνούμε από πλευράς εσωτερικής αγοράς αυτό είναι και το βασικό μας κήρυγμα, αν θέλετε, το βασικό μας μήνυμα. Ας το δείξουμε λοιπόν και στην καθημερινή μας ζωή. Άρα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή περιαγωγής σε σχέση με τις εγχώριες τιμές ε, των παρόχων και θα θέλαμε μηδενική προσέγγιση μέχρι το 2015 έτσι ώστε να μην μας πούν ε, οι παροχοί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τότε, θα φτάσουμε στη μηδενική βάση. Θα δούμε και τις εναλλακτικέ ως προς τις υπηρεσίες ε, περιαγωγής. Ποιες είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες, ε, τι γίνεται με το Wi-Fi, με τα δίκτυα Wi-Fi, έτσι ώστε και η περιαγωγή να γίνει πιο ανταγωνιστική. Θα προωθηθεί και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα της περιαγωγής και πιστεύω ότι αν υπάρχει ανταγωνισμός τότε όλα ε, βαίνουν καλώς για τον καταναλωτή στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει θα αναθεωρήσουμε τον κανονισμό περιαγωγής, σας το έχω υποσχεθεί αυτό, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του χρόνου. Αυτή είναι η τελική προθεσμία και θα επανέλθουμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τότε. Ε, ως προς την έρευνα και την καινοτομία, και όπως είπε ο κύριος Ρούμπιχ, Ο δημόσιος τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υποστηρίξει τις λεπικοινωνίες και τις, την πληροφορίες και την καινοτομία το ITC. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και σε αυτό το τομέα. Μιλώ για τη συνεργασία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρώπης. Αλλά μπορούμε να λάβουμε υπόψη και την από Ανατολή. Εάν συγκρίνουμε με ορισμένες χώρες της ε, από Ανατολής για να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σε εθνικό επίπεδο και σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Δεν πρέπει να αλληλοκατηγορούμεθα ότι δεν προωθούμε το ζήτημα παρκώς. Και όπως ξέρετε, επειδή ασχολείστε με το FP7, μιλάμε για μία αύξηση 16% μεταξύ 2010 ε, και 2013. Έτσι, να φτάσουμε, ώστε να φτάσουμε από 1,1 δισεκατομμύριο στο 1,7 το 2013. Έτσι ώστε να έχουμε ένα ετήσιο ρυθμό ε, αύξηση 4% που θα φτάσει μέχρι το διπλασιασμό. Θα πρέπει να γίνει η ίδια προσπάθεια από τα κράτη-μέλη, όπως είπε και το Συμβούλιο Ανταγωνισμό πέρσι το Δεκέμβριο. Όλοι είπατε, αλλά ιδιαίτερα ο κύριος ε, ε, Λάμπερτ κινήθηκε ιδιαίτερα προς το θέμα της στοχοθέτησης. Ίσως ε, ανέλαβα κινδύνους λόγω της ηλικία μου, γιατί δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή. Θα υπάρχει ένα βαθμολόγιο, γι' αυτό μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε πρόταση και με τις ε, κάρτες που σας έδωσα σας δείχνω ότι είμαι υπέρ της διαφάνειας και θα με στήσετε στον τοίχο αν δεν είμαι ιδιαίτερα αποδοτική. Άρα ανεξάρτητα από το ποιος επίτροπος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το έργο δεν είναι δική μου ψηφιακή ατζέντα, είναι της Κομισιόν. Και από εδώ και στο εξής είναι και του Συμβουλίου. Έχω πολλούς, υπάρχει μεγάλη συντροφικότητα, λοιπόν, και αν δεν τα καταφέρω δεν θα τα καταφέρω εγώ, σίγουρα θα ε, δεχτώ τις επικρίσεις όλων. Ελπίζω όμως στο τέλος της συζήτησης όλοι οι συνάδελφοι να συνεισφέρουν και το Συμβούλιο και εσείς ως Κοινοβούλιο. Για τα e-skills, για τις ε, ηλεκτρονικές δεξιότητες, έχει σημασία να υπάρχει ομοφωνία Γιατί κάποιος να επενδύσει σε έναν τομέα ε, αν δεν είναι σίγουρος ότι το τομέας αυτός θα τα καταφέρει. Εάν τα καταφέρουμε εμείς με την ψηφιακή ατζέντα και με την ψηφιακή κοινωνία, τότε θα διασφαλίσουμε τις 700.000 θέσεις. θα πρέπει να υπάρχει και ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός μεταξύ όλων αυτών. Άρα θα πρέπει και στο επόμενο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να ενταχθεί αυτό το σκέλος και να γνωρίζουν όλοι ότι καλό θα ήταν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να τους δώσουμε και τα κίνητρα. Δεν μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά ε, συγκρίνοντας με τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ταλαντούχους ε, επιχειρήσεις, με επιχειρήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μερικοί συνάδελφοι έφυγαν διότι είχαν άλλες υποχρεώσεις. Έχουμε οκτώ συναδέλφους που θα παρέμβουν. Επειδή και εγώ χρησιμοποίησα τόσο χρόνο, δεν μπορώ να σας ε, κάνω επικρίσεις, αλλά θα ήθελα να σας υποδείξω το ένα λεπτό παρέμβασης για να προχωρήσουμε σχετικά γρήγορα. Ε, ε, Τώρα, η κυρία Μερικίες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έλευσή σας εδώ κυρία Κρούς. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε και σας ευχαριστώ και για τους φιλόδοξους στόχους σας αλλά και τους φιλόδοξους στόχους του Συμβουλίου και οι δικοί μας πρέπει να είναι φιλόδοξοι. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που μίλησαν πριν από μένα ότι είναι ευκαιρία η τεχνολογία αυτή, ευκαιρία για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε σωστά τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως της ενέργειας, όπως της γύρανσης του πληθυσμού κτλ. Και βεβαίως να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη απασχόληση. Τώρα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δυνατότητα η ενέργεια, τι υποστήριξη δίνεται, θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην ε, Ολλανδία. Υπάρχει και η πρωτοβουλία Innovation Flex. Είχα την προηγούμενη εβδομάδα ευκαιρία να ε, συζητήσω με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην ICT και ε, υπάρχουν δυνατότητες να λάβει υποστήριξη ένα κεφάλαιο δηλαδή για να αρχίσει τις δραστηριότητε του. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι μπορούν να δοθούν για παράδειγμα κάποιες ε, εγγύσεις για να αρχίσουν ε, την δραστηριότητά τους. Ποιες είναι, τι σχέδια έχετε για παράδειγμα στον τομέα της υγείας όπου υπάρχουν Υπάρχει μεγάλη άγνοια πλευράς των ασθενών. Δεν θα έπρεπε να είναι καθήκον και των κυβερνήσεων να ε, προωθήσουν τις γνώσεις των ασθενών σχετικά με την ηλεκτρονική ε, υγεία. Τώρα, έχετε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πώς βλέπετε τις συνεχιζόμενες αυτές οι επαφές. Ε, μας υποβάλλατε την ε, ψηφιακή ατζέντα γρήγορα και σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσετε τις επαφές με τις ε, μικρές και μαζίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ και την κάρτα που διανύματε, την οποία βρίσκω εξαιρετική. Γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο ICT, την οποία είχατε, στην οποία συμμετάσχατε κι εσείς, μπορεί κανείς να ε, διαβάζοντας με το iPhone που ενδεχομένω διαθέτει μια κάρτα να έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ε, κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ την Επίτροπο που προσήλθε και μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε. Εγώ Πάντως θεωρώ πολύ ορθή την ψηφιακή ατζέντα. Ένα πρώτο θέμα είναι η υποδομή, broadband targets, στόχοι δηλαδή ευρέως φάσματος. Ε, και ευχαριστώ για την κάρτα αυτή, άλλωστε είναι ο πρώτος στόχος την οποία περιλαμβάνεται εδώ. Είναι σημαντικό να προωθηθεί η υποδομή ευρέως φάσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με το θέμα αυτό έχουμε ασχοληθεί και στα, και στα πλαίσια της δέσμη μέτρων τηλεπικοινωνιών. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κάνει ακόμα προτάσεις για τις επόμενες γενναίες συσκευών. Πάντως θυμίζω ότι το πακέτο τηλεπικοινωνιών έγινε δεκτό εδώ, έγινε, ενεκρίθη εδώ με μεγάλες πλειοψηφίες. Επίσης, σημαντικές πρέπει να είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα οπτικών ινών. Εγώ θα το τονίσω και τώρα, αλλά και σε κάθε συζήτηση που θα διεξαγάγω τα επόμενα δύο χρόνια μαζί σας, θα το θέτω το θέμα αυτό. Οι προϋπολογισμοί και στις 27 χώρες μέλη έχουν τα χάλια τους. Άρα χρειαζόμαστε την υποστήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε θέση και έχουν και την τεχνογνωσία, να προβούν σε επενδύσεις στα οπτικά δίκτυα πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να τις ενθαρρύνουμε, να τους χορηγήσουμε κίνητρα. Έχουμε ασχοληθεί με τα κίνητρα αυτά. Είπαμε ότι ο κίνδυνος των επενδύσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη. ή να υπάρξουν και δυνατότητες κοινών επενδύσεων. Περιμένω την ανακοίνωσή σας για το NGA. Δεύτερο, πολύ σύντομα. Όλοι συζητούν τώρα τις επιχειρηματικές πρακτικές τη Google. Τι, κάνει, τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τι θα κάνετε εσείς ως πρώην και ιδιαίτερα επιτυχημένη Επίτροπος του Αρμόδια για τον Ανταγωνισμό. Θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άποψη αυτή την περίπτωση Google. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Άκουσα προσεκτικά τι είπε σχετικά με τη δεύτερη αυτή ζωή της και για την πολιτική κατάσταση στις κάτω χώρες και για την ε, ψηφιακή ατζέντα για την οποία μας μιλήσατε και αναφερθήκατε σε ορισμένους τομείς. Εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα μιλήσατε για τα θέματα υγείας, τις φροντίδες υγείας και για αυτές μίλησε και η κυρία Μέρκης. Μιλούμε για benchmark, μιλούμε για ανταλλαγές. Αφενός η τεχνολογία λοιπόν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά είναι κατακαιρματισμένος ο κλάδος. Για παράδειγμα, Siemens και άλλε εταιρείε που έχουν ασχοληθεί πολύ με την ηλεκτρονική υγεία. Ορισμένες καινοτομίες έχουν καταλήξει στην αγορά, αλλά δεν προχωρούν τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυσκολίε, πολλά προβλήματα. Μιλήσατε για την επινοητικότητα, για τη δημιουργικότητα, αλλά τι μπορεί να κάνει κανεί συγκεκριμένα. Διατυπώνονται πολλοί στόχοι, αλλά στις χώρες μέλη ε, δεν προχωρούν τα πράγματα, διότι οι πόροι είναι όλο και πιο περιορισμένοι. Εάν δεν διατυπώσουμε μια κοινή ατζέντα, οριζόντια, θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Αλλά πάντως η οριζόντια διάσταση δεν είναι επαρκής. Χρειάζεται να εξετάσουμε και την κάθετη διάσταση. Επένδυση λοιπόν στην έρευνα είναι σημαντική για όλες τις ε, χώρες μέλη και να φροντίσουμε ώστε τα σχετικά προγράμματα να ε, προωθηθούν και στο εθνικό επίπεδο. Όπως είπε και η κυρία Μέρκες, θεωρώ και εγώ ότι συχνά γίνονται επενδύσει στη βάση από δημόσιες επιδοτήσεις δηλαδή, δίνονται εγγύησεις και τελικά νομίζω ότι πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι καινοτομίε αυτές ε, να συγκεκριμενοποιούνται. Δεύτερο σχόλιο. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι και ενήλικοι στα κοινωνικά δίκτυα και ιδίω για τους νέους είναι σημαντικό, είναι θέμα και εμπιστοσύνη δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που δεν τηρούνται οι κανόνες, αναγκαστικά αυτό οδηγεί σε προβλήματα. <clears throat> Αναφέρατε ορισμένα δεδομένα. Μέχρι τώρα όμως, ό,τι αφορά την προστασία, την ασφάλεια, νομίζω ότι δεν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα. Σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω να τηρείτε το χρόνο σας. Λυπούμε πολύ, αλλά έτσι είναι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για την εισήγησή της, γιατί όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για να παρακολουθήσουμε αυτές τις στοχοθετήσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που μου δώσατε στις 27 Μαΐου σε μία γραπτή μου ερώτηση για την επιδείνωση στην κατάσταση των ΜΜΕ εν ώψη της ε, χρηματοοικονομικής ε, κρίσης και σε σχέση με την ελεύθερη πληροφόρηση και έκφραση των ε, πολιτών. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια δύσκολη θέση. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε οπωσδήποτε την ε, ψηφιακή ατζέντα και να δούμε και τις κοινωνικο καταστάσεις τις οποίες δεν είχαμε συναντήσει μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτός ο εξυγχρονισμός της ψηφιακής ατζέντα. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών που γνωρίζουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική ύφεση και που δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους για να εξυγχρονίσουν αυτό το πλαίσιο. Και υπάρχουν και επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την οικονομική κρίση, όπως για παράδειγμα ο τύπος, ο ημερήσιος τύπος. Πώς βλέπετε αυτή τη μετάβαση του γραπτού ημερήσιου τύπου στην ψηφιακή ατζέντα πώς μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί χάρτου, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε εθνικό επίπεδο, διότι υπάρχουν και οι οικονομικές, μάλλον κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή ατζέντα ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν μάθει και προτιμούν να διαβάζουν μια ε, εφημερίδα επί χάρτου και δεν θέλουν να προσφύγουν σε ψηφιακά μέσα. Εσείς μου είπατε στην απάντηση ότι τη στιγμή που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν τομέα που αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες και ο οποίος είναι κατεξοχήν ιδιωτικός και τι εγγυήσει ανεξαρτησίας υπάρχουν στην ελεύθερη έκφραση σε αυτή την περίπτωση τη στιγμή που θα εξαρτώμαστε από την ελεημοσύνη της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι θα γίνει μια άλλη συζήτηση μετά από αυτήν. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να είσαστε σύντομοι στις ερωτήσεις. Θα προτείνω οι τέσσερις τελευταίες ερωτήσεις να υποβληθούν τώρα και να απαντήσει συνολικά η Επίτροπος στις ερωτήσεις, έτσι ώστε να τις ε, ομαδοποιήσει όπως κρίνει καλύτερα, θεματικά μάλλον, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο μας. Σας παρακαλώ για τους τέσσερις ομιλητές να είσαστε σύντομοι. Η κυρία Τσικάου, and uh, uh, um, Τσικάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να αρχίσω ρωτώντας πώς έχει το πρόγραμμα κάλυψης 100% της ευρυζωνικότητας. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά σχέδια οικονομικής ανάκαμψης υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να δοθούν μέχρι το 2000, στο τέλος, μέχρι το του 2010 για να καλύψουμε κατά 100 της 100 την ευρυζωνικότητα. Θα ήθελα όμως να μας πείτε από πού ξεκινάμε για αυτό το στόχο. Ως προς το πρόγραμμα ΕΝΙΣΑ εγώ είμαι υπέρ της ε, διεύρυνσης της θητείας, της εντολής αυτής, ιδιαίτερα ως προς ορισμένες εκτελεστικές δυνατότητες της ΕΝΙΣΑ για να αντιμετωπίσουμε θέματα κατεπήγοντας, γνωρίζοντας ότι το ICT είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή επικοινωνία, τεχνολογία και καινοτομίες. Τι γίνεται ως προς τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται και διασυνοριακή διαλειτουργικότητα αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν το 16% του ΑΕΠ Υπάρχει δήλωση του Μάντσεστερ που ορίζει ότι το, μέχρι το 2015 το 15% όλων των δημοσίων αγορών θα γίνεται μέσω e-procurement και τι θα κάνετε με την τιμολόγηση, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό invoicing έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση ως προς την ε, διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών, θα ήθελα να μας πείτε τι θα γίνει με την επικύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Και το τελευταίο είναι το εξής. Στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ζητήσει τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν αν δεν την έχουν, μία στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας, γιατί με την ευρυζωνικότητα και με την κάλυψη 100% και λόγω ηλεκτρονικών προμηθειών θα πρέπει να προβάλλουμε μία στρατηγική κυβερνοασφάλειας και μέσα στον ευρυζωνικό χώρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ η κυρία Κορλάνσκα Μποβίνσκα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτούς τους ε, φιλόδοξους στόχους γιατί είναι απόλυτα σαφής και θα πρέπει ε, κάθε χρόνο να λαμβάνουμε από σας μια τέτοια καρτέλα με πληροφορίες για την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτών των στόχων. Σε σχέση με τους στόχους μιλάμε για 100% ε, χρήσης του διαδικτύου μέσα στα πλαίσια της ευρυζωνικότητας και το άλλο είναι η ταχύτητα ε, παροχής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους γιατί υπάρχουν ε, χώρες που βρίσκονται πολύ, σε πολύ καλό δρόμο στην ευρυζωνικότητα ενώ άλλες, ενώ άλλες χώρες υπολείπονται αυτής. Τι θα κάνουμε με τις χώρες που έχουν μείνει πίσω. Μιλήσατε για συνεργασία με κυβερνήσεις. Πώς θα ε, τα βλέπετε τα πράγματα. Ε, λυπάμαι που πρέπει να φύγω γιατί θα πρέπει να μιλήσω σε άλλη επιτροπή, αλλά η Αντζέλικα θα μου πει τι, τι μου απαντήσατε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ροντή. Ευχαριστώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλήρους αποτυχίας, διότι πια αποδοτικές ε, υπηρεσίες δεν τα καταφέρνουν ούτε τον καλλιλέο ούτε το ΊΤΕΡ. Εσείς μας μιλάτε για ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες, μα έχουν κουραστεί πλέον οι πολίτες για, με όλες αυτές τις υποσχέσεις. Πιστεύω ότι η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα είναι κάτι το πολύ βασικό. Πώς θα τηρήσετε τις υποσχέσεις σας τόσο γρήγορα μπορείτε να μας δώσετε εγγυήσεις και επίσης το περιεχόμενο δεν θα φύγει θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία δεδομένων, καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας, πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια και αποπτία του περιεχομένου. Κύριε Φόλ, που είσαστε και τελευταία. Λυπούμε που δεν ήμουν εγκαίρος εδώ γιατί συναντήθηκα με τον Υπουργό της χώρας μου για θέματα παρόμοια με τα δικά σας και δείχνει τη σημασία που δίνει η χώρα μου. Τώρα, για το ευρύ φάσμα βλέπω ένα είδος ε, πολιτών δεύτερης κατηγορίας, αυτοί που δεν έχουν δηλαδή. Στην ε, περιοχή μου βλέπω πολλές καινοτόμες λύσεις από διάφορες επιχειρήσεις για να προωθηθούν τα δίκτυα αυτά και στις ε, περιοχές της Υπέθρου. Όμως να εξευρεθούν χρήματα είναι δύσκολο για την ώρα. Είναι λοιπόν σημαντικό να βελτιστοποιήσουμε τις υφιστάμενες υποδομές για παράδειγμα για τα σχολεία να έχουν ε, τέτοια διασύνδεση τα παιδιά. Έχουν καμιά φορά, αλλά όταν πάνε σπίτια τους στα χωριά δεν έχουν. Εδώ λοιπόν ε, είναι σωστό να, μπορεί, να μπορούν να διασυνδεθούν με την υποδομή του δημόσιου τομέα. Τώρα, υπάρχει και μεγάλη σύγχυση σχετικά με τις ε, ενισχύσεις που δίνει η κοινότητα, παρόλες τις δηλώσεις του περσινού χρόνου. Παρότι λοιπόν προσπαθήσατε να διευκρινίσετε τα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα μπορούσε ο δημόσιος τομέας να ε, βοηθήσει στην κάλυψη των κενών, των περιοχών εκείνων που βρίσκονται ακόμα σχετικά πίσω. Είναι λοιπόν περίπλοκα τα πράγματα, πρέπει να, γίνουν, να ληφθούν μέτρα για να ε, βελτιωθούν και να απλοποιηθούν τα πράγματα αυτά. Ε, αντιδράσω σε αυτά που είπε η κυρία Φολ. Εάν υπάρχουν ε, ερωτηματικά, να με ρωτάτε πώς, από ποιον και γιατί. Διότι γίνεται χρήση αυτών των επιχειρημάτων από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, δεν μιλώ για σας. Εσείς είπατε ότι δεν πρέπει να υπάρξει μία χαμένη, χαμένη γενιά και δεν θα πρέπει να υπάρχει χαμηλή προσδοκιμότητα στην ε, κάρτα. Είναι απόλυτα σαφές, ε, το 2013 θα μπορεί όλη η Ευρώπη να είναι ε, ψηφιακή. και θα μπορέσετε να το δείτε, δεν υπάρχει ε, αμφιβολία, αλλά θα πρέπει να δεσμευτεί το Συμβούλιο διότι αυτός είναι ο, σημαντικός, ο βασικός μας συνομιλητής. Μιλάμε για αγροτικές περιοχές, μιλάμε για όλους. Και νομίζω ότι σας το εξήγησε και ο αντιπρόεδρο, η αντιπρόεδρό σας. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας ε, στο διαδίκτυο. Δεν μιλάμε για καλωδιακή, πρόσβαση οπτικές ίνες. Θα πρέπει όλα αυτά να φτάσουν και στις αγροτικές περιοχές. Ε, εάν ε, αναθεωρηθούν οι κρατικές επιδοτήσεις και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί και ο πρόεδρος Μπαρόζο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Εάν κάτι δεν είναι σαφές να μου το κοινοποιείτε. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σαφές, αλλά αυτό που με φοβίζει είναι ότι στο, στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, στην προηγούμενη μάλλον θητεία της Κομισιόν, μιλήσατε για ένα δις ευρώ. Είναι δύο δις τα χρήματα αυτά που είχαν προγραμματιστεί. Και είχαμε πει ότι θα δαπανηθούν για την ευρυζωνικότητα και μόνο το εν τρίτον τελικά δαπανήθηκε για την ευρυζωνικότητα. Τα άλλα θέματα αφορούσαν καταναλωτικές δαπάνες. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Ή θα είμαστε σαφείς Ω ως προς την κατεύθυνση αυτή του ψηφιακού μέλλοντος, αλλά τότε δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με προεκλογικά ζητήματα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται χρόνος πριν αποδώσει μία επένδυση στον ψηφιακό κόσμο για να δείξουμε σε όλους ότι πρόκειται για την απασχόληση, για την οικονομία, για μια κοινωνική στάση των ανθρώπων. Θα πρέπει να είμαστε επικοινωνιακοί ως προς όλα αυτά. Θα είμαι ιδιαίτερη, ιδιαίτερα σύντομη. Κλιματικές αλλαγές. Η κυρία Μαρκής το έθιξε αυτό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να το εντάξουμε και στις ε, κλιματικές ε, αλλαγές. Θα πρέπει να έχουμε ένα ευφυές δίκτυο για να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί ως προς αυτό. Θα συνεργαστούμε με τη βιομηχανία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορώ να υποχρεώσω μία κυβέρνηση να το δεχτεί, αλλά μπορώ να το προβάλλω, να πω ότι θα ήταν συνετό να ακολουθήσει αυτή την πολιτική μία κυβέρνηση. Για να έχουμε μία κατάσταση ολικού κέρδους. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφής. Εμείς, σαν ευρωπαϊκή βιομηχανία, θέλουμε να δούμε ε, το εξής. Όταν χρησιμοποιούμε ένα, έναν ε, ε μετρητή, δεν το κάνουμε μόνο για το κλίμα, αλλά είναι επικερδές γενικότερα, δηλαδή είναι ένα λιγότερο δαπανηρό σύστημα και συμφέρει. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς ε, το διαδίκτυο. Το άλλο θέμα που θίξατε είναι ύψης της σημασίας ε, για μας. Είναι μεγάλη ε, δυνατότητα και ευκαιρία για μας. Ε, πρότεινα διάφορες δράσεις, ξεκινώντας από τον εξοπλισμό για την πρόσβαση online και σε έναν κατάλογο διαλειτουργικότητας και σε επίπεδο νοσοκομείων και ασθενών. Θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να ταξιδεύει με το σπίτι του, με άλλα λόγια. Γιατί πολλές φορές δεν αντιτάσσονται οι άνθρωποι σε αυτές τις νέες ευκαιρίες, αλλά αυτοί που φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επιβλαβές για τη δραστηριότητά τους, ας πούμε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ούτω καθεξής. Άρα χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων. Η κυρία Νίμπλερ ε, μίλησε για την ε, γενικότερη στρατηγική. Έχουμε προβάλει τις κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών ε, επιδοτήσεων ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα NPAs, δεν μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το πλαίσιο ολοκληρωτικά και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να υποσκάψει την ανταγωνιστικότητά μας και την οικονομική ανάκαμψη. Άρα θα πρέπει να έχουμε συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αξίζει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό θα ήταν επικερδές γενικότερα. θα ήθελα να κινηθούμε προς ένα πιο ε, επικοδομητικό τρόπο. Ως προς το Google τώρα. Ο συνάδελφος Αλμούνια το ερευνά ε, αυτό το θέμα της συμπεριφοράς του Google, αλλά είναι πολύ ε, πρόωρο να σας ανακοινώσω οποιαδήποτε μέτρα. θα πρέπει να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό Google κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ε, συνάδει με τη δράση του κυρίου Αλμούνια. Γνωρίζω το ε, θέμα που θίξατε. Θα αναφερθώ και στην προγενέστερη γραπτή απάντηση που σας έδωσα η ευρυζωνικότητα και οι επενδύσεις απάντησα και είπα ότι θα πρέπει να συμβαδίζουμε όλοι. Δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει μια επένδυση στην ευρυζωνικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και ως προς την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή, η οδηγία του 99 ορίζει την ηλεκτρονική υπογραφή που θα αποτελεί μέθοδο ταυτοποίησης και αυτή η υπογραφή είναι αναγνωρίσιμη. Βρισκόμαστε σε ένα εμβριακό στάδιο αναγνωρισιμότητας θα πρέπει να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης και για την ε, ταυτοποίηση και θα το αναθεωρήσουμε αυτή την οδηγία του 99. Είναι αρκετά παροχημένη. Προς την ερώτηση, ως προς την κυρία Κουλάνσκα την ερώτηση της. Όταν ασχοληθώ με την στρατηγική ευρυζωνικότητα, θα ασχοληθώ και με τη χαρτογράφηση αυτή και το συντονισμό μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και θα δούμε τι θα κάνουμε και με το θέμα του φάσματος. Όλα αυτά θα σας τα κοινοποιήσω το ταχύτερο δυνατόν. Μίλησα για την ευρυζωνικότητα, προτείνουμε μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει ε, και πρόσβαση στο περιεχόμενο, να διευκολυνθεί και βεβαίως να είναι και νόμιμη. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τα επόμενα πέντε χρόνια, μίλησα για τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων την ε, λογοδοσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρχει και διασυναριακότητα και δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων. Και αυτό αφορά και την ε, οριζόντια ολοκλήρωση διαχείρισης. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και για τον έξτρα χρόνο που μας διαθέσατε. Είμαι βέβαια ότι και στο μέλλον θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε και ότι τώρα πρόκειται απλώς για μια αρχή. Σας ευχαριστούμε.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 Αγαπητοί νύχοι, στις 18 2009 ε, η Κομισιόν μας δίδασε μια ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα για το διαδίκτυο. Αναθέσαμε την έκθεση στον Φρανσίσκο Ζουζά Βάγνερ. Θα το συζητήσουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο και στις 15 Ιουνίου θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ο εισηγητής για αμέσως το λόγο. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να καθησυχάσω τα μέλη της Επιτροπής, τονίζοντας ότι θα είμαι σύντομος γιατί είχαμε ένα ε, πολύ μεγάλο απόγευμα. Ε, σχοληθήκαμε με θέματα και αυτής της έκθεσης και νομίζω ότι έχουμε μία σαφή ιδέα για το τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Επιπροσθέτως θα ήθελα να ευχαριστήσω, πριν μπω στην αιτιολογική σκέψη, θα ήθελα να ευχαριστήσω του Σκιώδης για τη συνεργασία, για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Με τους Σκιώδης και με τις τροπολογίες ε, διορθώθηκαν πολλά για να βελτιωθεί το αρχικό κείμενο. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τις τροπολογίες που θα δούμε και αύριο. Υπάρχουν πέντε ομάδες τροπολογιών. Η πρώτη αφορά το διαδίκτυο ως δημόσιο αγαθό. Είναι ε, η αρχική διατύπωση της έκθεσής μου και εδώ, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα δημόσιο κοινό αγαθό, λέμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Η δύο αφορά ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό αποτέλεσε μεγάλη, μέρος μιας μεγαλύτερης ε, ευρύτερης συζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι οι αξίες αυτές εξασφαλίζονται. Δηλαδή να τις υπερασπιζόμαστε σε όλα τα διεθνή φόρα. Ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του και την προάσπιση αυτών των αξιών και δικαιωμάτων στα φόρα εκείνα όπου συμμετέχουν χώρες που δεν συμμερίζονται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μας ενισχύσει και να ενισχύσει και τις αξίες μας. Πρόκειται για αξίες του πολιτισμού μας και επιμένουμε για αυτές. Η τρίτη τροπολογία αφορά τους ε, περιορισμούς στην χρήση και πρόσβαση. Τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί για την προστασία των μικρών παιδιών και για την καταπολέμηση της παιδικής περνογραφίας. Εδώ μιλάμε για δύο βασικές αρχές, την αρχή της αποτελεσματικότητας και την αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται για δύο αρχές που συνυπολογίζονται ε, στη συνθήκη, όπως ορίζει και επεξηγεί και το ΔΕΚ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της έκθεσης. Η τροπολογία υπαριθμών 4 μιλά για επιπρόσθετες αρχές που θα πρέπει να ενταχθούν στο κείμενο. Μιλάμε για βασικές αρχές, όπως μας είπε και η Επίτροπος, δηλαδή η αρχή της πολυπλευρικότητας, διαλειτουργικότητας, ουδετερότητας του δικτύου, της ευθύνης του ιδιωτικού τομέα που ασχολείται καθημερινά με το θέμα Όλες αυτές οι αρχές μας απασχόλησαν εδώ όλο το απόγευμα. Γι' αυτό μιλάμε για την τροπολογία συμβιβασμού Υπάρχουν 4. Επίσης θα θέλαμε να επιμείνουμε στο συντονισμό, στο θεσμικό συντονισμό σε όλα τα χώρα του διαδικτύου. διότι δεν μιλάμε μόνο για το ΙΚΑΝ, αλλά και για άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις. Ήδη στην αρχική μου έκθεση τονίζουμε την ε, ανάγκη συντονισμού όλων των ε, θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών στην διαχείριση και διακυβέρνηση του διαδικτύου. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους της έκθεσης. γιατί οι επικρίσεις που απευθύνονται σε εμάς για το γνώσο ότι ε, δεν λειτουργούμε εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν. Να ορίσουμε δηλαδή κοινέ θέσεις από το θεσμικό μας πλαίσιο, κομισιόν, συμβούλιο κλπ. Για να δούμε πώς διαχειριζόμαστε το ίντερνετ. Και θα εντάξουμε και ορισμένες ε, βελτιώσεις για έναν εναλλακτικό μηχανισμό διαιτησίας με βάση το ΙΚΑΝ και μία εναλλακτική χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, καθοριστικός επηρεασμός της δραστηριότητας του ΙΚΑΝ και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη του ΙΚΑΝ να προέρχονται από, όλο τον κόσμο, από όλες τις περιφέρειες. για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του πλαισίου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και θα ήθελα να υποστηρίξετε όλες τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού. σε θέματα ίσονος ε, σημασίας δεν επιμένουμε, διότι εντάσσονται αυτά τα, τα στοιχεία στην έκθεση και από τις αρχικές ε, τροπολογίες. Και αυτό που έχει σημασία είναι η διατύπωση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επί του θέματος. Διαβάσαμε την έκθεση της ΛΥΜΠΕ και θα την αναλύσουμε ακόμα περισσότερα, αλλά συμφωνούμε με την διατύπωση όπως ορίστηκε σήμερα το απόγευμα. Με αυτά έχω να σας πω και περιμένω τις δικές σας υποδείξεις. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Βάντσον. Voorzitter, ik kan even kort als eh, de, de presentatie van onze... ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή μας γιατί παρουσίασε τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Είχαμε ήδη μία ανταλλαγή απόψεων δύο φορές. Τώρα ο εισηγητής σχολίασε της ε, τροπολογίες, αλλά θα πρέπει βέβαια οι συμβαστικές τροπολογίες να αντικαταπτύσσουν την ισορροπία που έχει επιτευχθεί. Ε, αυτό που έχουμε πετύχει θα πρέπει να εκφράζεται ξεκάθαρα στο κείμενο και να λέγεται πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει διάκριση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Δεύτερον, Πρώτα κάτι που έφτασε αρκετά αργά, η γνωμοδότηση δηλαδή της ε, Νομικής Επιτροπής. Την εξετάσαμε στη δική μας ε, πολιτική ομάδα. Εσείς λέτε ότι σε γενικέ γραμμέ μπορείτε να συμφωνήσετε. Εγώ έχω μία πρόταση να κάνω για την παράγραφο 6 όπου αναφέρεται ζητεί από τις κυβερνήσεις να αποφεύγουν την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο με μέτρα λογοκρισίας, διαλογής, περιεχομένου, παρακολούθησης ή άλλα. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη διαλογή του περιεχόμενου αυτού καθεαυτού. Αυτό δεν είναι ε, πλήγμα προς την ιδιωτική ζωή. Αλλά ο όρος παρακολούθηση, monitoring, θα μπορούσε να διαγραφεί, αλλά δεν θα είναι αυτοβελτίωση Θέλουμε λοιπόν κατά τμήματα ψηφοφορία για αύριο. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Κατρίν Τροτμάν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή μας που πολύ καλά πρόθεσε τις ε, συμβαστικές αυτές με την οποία, τις οποίες μπορώ να σας πω ότι συμφωνεί η ομάδα μας γιατί μπορέσαμε να τις εξετάσουμε στην ε, προπασκευαστική μας ε, συνεδρίαση εργασίας και πέτυχε νομίζω τις διατυπώσεις που ικανοποιούν και επιτρέπουν να μειωθεί ο αριθμός των τροπολογιών κατά κάποιον τρόπο, πράγμα που είναι πάντα πολύ χρήσιμο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή γιατί τώρα που προετοιμάζουμε το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Και νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το έτοιμά μας ε, για μια αντιπροσωπεία στο πέμπτο αυτό φόρουμ πιο σημαντική από εκείνη που είχαμε στο παρελθόν και που γίνεται στο Βίλνιο, στη Λιθουανία και το κοινοβούλιο μας θα μπορούσε να οργανώσει ένα εργαστήριο πάνω στην έξω του Σώσα Βάκνερ. Δηλαδή πολυγλωσία και ταυτόχρονα πολυμορφία της έκφρασης. Έχουμε λοιπόν βασικές αναφορές εδώ. Έχουμε ένα κείμενο το οποίο διευκρινίζει τα πράγματα πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις επιμέρους αρμοδιότητες για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου μας ανοίγει μελλοντικές ε, προοπτικές, είναι ακριβές, ε, σαφές, ε, ενθαρρυντικό για την εξέλιξη του ΕΚΑΝ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή έκθεση και θα χαρούμε αύριο να μπορέσουμε να εκφραστούμε έτσι ώστε να κατανοήσω ότι αυτή είναι η στάση ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ο Φιπλάμπα έχει το λόγο. Ναι, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Όχι γενική, αλλά διαδικαστική μάλλον. Γιατί πάλι όταν συζητάμε για την προστασία των παιδιών, ανοίγουμε τη συζήτηση για το πώς θα μπορούν να γίνουν αυτοί οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και αυτό εμένα με ενοχλεί, γιατί διαπραγματευθήκαμε ένα προβιβασμό μέσα στα πλαίσια της τρίτης ανάγνωσης ε, της ΔΕΜΣΕΚΟΜ. Γιατί πρέπει να το ανοίξουμε, θέλουμε να πούμε τα ίδια πράγματα, δεν υπάρχει κανένα Είναι παράδοση του σώματος να προσπαθήσει σε κάθε έκθεση που κάνουμε να καλύπτουμε τα πάντα. Αλλά νομίζω αυτό οδηγεί σε σύγχυση, γιατί έτσι υπάρχουν αντιφάσεις ε, μεταξύ των διαφόρων κειμένων. Αυτά έχω να πω. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την Κατρίν και να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έκανε ένα έργο πραγματικό μέσα σε πολύ συμβιωτικό και συνεργάσιμο πνεύμα. Αλλά θα ήθελα να είμαστε λιγότερο αμφιβολεγόμενοι μέσα στα κείμενα και να μην επαναλαμβάνουμε τα πάντα, γιατί αυτό δεν ικανοποιεί όλους. σε ευχαριστώ, δεν βλέπω κανένα λόγο να θέλει το λόγο. Α, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Σας Γκοστέτ, παρακαλώ. Ναι. Δεν είχα ζητήσει προηγουμένω το λόγο. Δεν μπορείτε να ξέρετε ότι το ζητούσα τώρα. Με δύο λόγια θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτού του τύπου τα κείμενα και να μην επανερχόμαστε συνεχώς στο δέσμι τηλεκομ, Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε να πετύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των παραγωγών και τη διασφάλιση των βασικών μας δικαιωμάτων. Να βρούμε λοιπόν εκεί τη σωστή ισορροπία και φοβούμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν αποκλήσει μέσω της οδηγία αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τώρα πράγματι δεν βλέπω κάποιον άλλο βουλευτή να ζητάει το λόγο. Ο κ. Δίπελ τη ε, Κλασική Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιό χαιρετίζει την έκθεση αυτή και αυτή την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση και συμμεριζόμαστε αυτά που είπε ο Συγητή για το διαδίκτυο σαν ένα κοινό αγαθό της ε, κοινέ ε, ευρωπαϊκέ αξίε που θέλουμε να προωθήσουμε και την ανάγκη να υπάρχει μία φωνή μόνο με την οποία θα μιλάει η Ένωση. Επίσης εκτιμούμε το γεγονός ότι εκφράζεται τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την καταπολέμηση του εγκλήματος στο κυβερνόχωρο και τα θεωρείται τα πιο σημαντικά θέματα. Όσον αφορά την εμπλοκή τους, ε, των θεσμικών οργανωσίων στο ΕΚΟΝ, ε, πιστεύουμε ότι αυτή η κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή είναι μία από τι επιλογέ, όχι η μόνη. Και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη αξία στην πρόταση να μειωθούν τα φιλοαγόμενα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να μπορούμε να έχουμε μία αναθεώρηση εξωτερική για να είναι ανεξάρτητη. Έχει αναφέρεται επίση η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα διεθνού κοινότητα και να μπορέσουμε έτσι να προτάσουμε το ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτηση με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νίβερ. Πρώτο ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Ήθελα επίση την προσοχή του σε ένα πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε για την θέση της ε, νομικής επιτροπής όπως στην παράδειγμα 8 προτείνει μία σειρά σκέψεων που αναφέρονται αλλού εκτός από τα, ε, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Μήπω θέλει ο να αναφέρει κάτι τέτοιο ο, μέσα στα πλαίσια τη διακυβέρνηση του δικτύου, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μου λέει η γραμματεία ότι η τροπολογία 8 της νομικής επιτροπή δεν ψηφίστηκε γιατί ήταν καλυμμένη. Ναι, είναι καλυμμένη για όλα τα άλλα, αλλά όχι για τα ευρωματικά δικαιώματα. Τι έχει να πει ο εισηγητής από αυτό. Vamos a Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις παρατηρήσεις ξεκινώντας από τον κύριο Βαν Νίστελ Ρόι για να του πω ότι πράγματι Η, έκθεση της ΛΥΜΠΕ ήρθε εδώ και πολύ λίγο χρόνο, τη λάβαμε εδώ και πολύ λίγο χρόνο σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να τη διαβάσουμε και να λάβουμε θέση. Βεβαίως ε, μας πιέζει ο χρόνος ε, διότι θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο και η Λίμπε μας έδωσε το κείμενο την τελευταία στιγμή. Και δεύτερον, σε σχέση με την κυρία Τράουτμαν θα ήθελα να την ευχαριστήσω Νομίζω ότι πράγματι αυτή η έκθεση μπορεί, είναι χρήσιμη για να ενδυναμώσει τη θέση του Κοινοβουλίου σε αυτά τα φόρα. Και αυτός είναι ένας από τους ε, βασικούς μας στόχους στο εγγύς μέλλον. Και όπως μας είπανε και ο, σινιόρ, και ο κύριος Λάμπερτ, με συγχωρείτε, και η κυρία Γκρόστετ, με αυτό το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Λάμπερτ και με την κυρία Γκροστέτ, γιατί από την πρώτη φορά που ε, παρεμβήκαμε επί του θέματος, τόνισα ότι το θέμα του διαδικτύου είναι ένα θέμα ευρύτατο και ιδιαίτερα περίπλοκο. Και εμείς δεν μπορούμε να θίξουμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που βρίσκονται σε αυτή τη μεγάλη κοιλιά, ας το πω έτσι, που είναι το ίντερνετ. Άρα, μιλάμε για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, όπως μας το όρισε ε, η Κομισιόν. Μιλάμε δηλαδή για έναν απέραντο κόσμο. Μιλάμε για το πακέτο Telecom το οποίο ήδη ψηφίστηκε και θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τους ε, σκιώδεις να περιορίσουμε κάπως το θέμα ως προς τη διακυβέρνηση, διαχείριση και ούτω καθεξής. Όμως, ανέκυψαν και άλλα ζητήματα στο μεταξύ και γι' αυτό και ανακύπτουν και επιμέρους ζητήματα, τα δικαιώματα των ανηλίκων, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως αυτό το θέμα έχει ενταχθεί, αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας τώρα δηλαδή διαδικαστικά βρισκόμαστε στο τέλος του κεφαλαίου αυτού. Αυτή είναι η δική μου θέση. Επιμένω γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε τα πάντα παντού. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο και δημιουργεί μεγάλη σύγχυση. Γιατί διαβάζουν τα κείμενά μας και εκτός θεσμικών οργάνων. Και αυτό ακριβώς λέω και στους συναδέλφους που επιμένουν, ότι θα πρέπει να βάζουμε όρια στα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ και εκεί. Δεν είναι απεριόριστα, ούτε μπορούν να είναι. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Τι έχετε να πείτε. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια μισή εφαρμογή αυτού που είπα. Θέλω ακόμα να προσθεθούν διάφορα θέματα σε μια έκθεση. Δεν λέω ότι είναι τελείως άσχετο, αλλά κοιτάξτε το θέμα των μορφωτικών δικαιωμάτων είναι αρκετά ευρύ και να το ξαναβάλουμε έτσι από το παραθυράκι την τελευταία στιγμή σε αυτή την έκθεση δεν είναι σωστό και θα ήταν καλύτερα να το αποφύγουμε. Δεν λέμε την τελευταία λέξη εδώ, ούτε η τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο θα έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων. Α μην δοκιμάσουμε εδώ να δημιουργήσουμε έτσι ένα τετελεσμένο γεγονός προσθέτοντας έτσι τα γλίγορα τρεις λέξεις μια έκθεση. Μα με συγχωρείτε, δεν πρόκειται για να προσθέσουμε στα γλίγορα ε, τρεις λέξεις, αλλά απλώς θέλουμε να λάβουμε υπόψη την τροπολογία της νομικής επιτροπής που νόμιζε η γραμματεία ότι είχε καλυφθεί αυτό, αλλά δεν ήταν καλυμμένο. Νομικά θα πρέπει νομίζω να το προσθέσουμε. Μα το λέτε η γραμματεία έκανε ένα σφάλμα και θέλουμε να το διορθώσουμε. Τι να σας πω, τότε ας πάρει μια άλλη θέση η γραμματεία. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Δεν είναι ότι έσφαλε η γραμματεία. Είναι ότι η γραμματεία θεώρησε, καλός ή κακός, ότι το σύνολο κάλυπτε το επιμέρους. Ότι όταν μιλάμε για βασικά δικαιώματα, γενικά, το γεγονός το ότι αναφέρουμε ένα από αυτά, δηλαδή τα δικαιώματα βηματικής ιδιοκτησίας, τυπικά δεν προσθέτει τίποτα. Μπορούμε να το ζητήσουμε εδώ. Αυτή είναι η θέση του κυρίου Ντί. Με τελευταία αναλύση, ο πρόεδρος αύριο θα πρέπει να βρει τη λύση. Εγώ αυτό που είπα στον κύριο Ντί ήταν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα κατά πόσον ο εισηγητής δεχόταν να εντάξει αυτό το στοιχείο σε κάποιο άλλο τμήμα της έκθεση του. Οποία αναφορά αυτή θα είχε νόημα. Εντάξει. Εδώ συμφωνώ με τη θέση της γραμματείας ότι άμα αναφέρουμε ένα βασικό δικαίωμα, μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Λοιπόν, εμείς επιμείνουμε σε αυτή τη θέση της γραμματείας. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα βασικά δικαιώματα, δηλαδή η καταπολέμηση διακρίσεων, ρατσισμός, ξενοφοβία κλπ. Δεν είναι βασικό δικαίωμα το δικαίωμα τη πνευματική ιδιοκτησία, το είναι ένα δικαίωμα που δημιουργούνται με μια πολιτική απόφαση. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αφορά στα βασικά δικαιώματα και τα πνευματικά δικαιώματα είναι πολιτική απόφαση. Και η νομική επιτροπή μας το πρότεινε στη δική μας επιτροπή. Αυτό ήταν. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος θα πρέπει να βρει τη λύση. Α, ωραία. Εντάξει. Ας βρει ο πρόεδρος τη λύση. Αύριο. Παρακαλώ. Τολμώ να επιμείνω, γιατί αυτό το θέμα δεν το είδαμε. Συμφωνώ με αυτά που μόλις είπε ο Πρόεδρος. Άλλο τα θεμελιώδη δικαιώματα και άλλα τα θέματα κοινή νομοθεσίας. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ένα συγκεκριμένο θέμα περνάει, μπορεί να περάσει ή όχι στην αυριανή ψηφοφορία. Κατανοεί ο Πρόεδρος ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να, θα πρέπει να ψηφιστεί. Δηλαδή, αν θέλετε όμως εσείς ντε και καλά να ψηφιστεί, εγώ αντιτίθεμαι. Εάν ήθελα να ενταχθεί στο κείμενο, θα το είχα κάνει εδώ και πολύ χρόνο, για τους λόγους που σας εξέθεσα. <coughs> βασίζομαι στην ε, καλή διαχείριση του Προέδρου και της Γραμματείας. Euh, Ωραία, άρα θα το δούμε αύριο. Άρα η γνωμοδότηση ΛΥΜΠΕ θα αλλάξει τον ε, κατάλογο ψηφοφοριών. Άρα οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αλλάξουν τη θέση τους. Θέλετε να πείτε κάτι. Zoals eh, de voorbereiding van de stemming is dat wij zeg maar, als EVP vragen om ons... Για την eh, προετοιμασία, εμείς ως ΕΛΚ θα ζητήσουμε ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτό το κομμάτι και το υπόλοιπο θα το ορίσει ο εισηγητής. Πρόταση, η πρότασή του μας βρίσκει σύμφωνος επί του παρόντος. Σας ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν. Στα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, διακόπτουμε τη συνεδρία. Θα συνεχίσω αύριο στι 9.